Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Κυρίες και κύριοι, λέει ο Πρόεδρος, καλημέρα. Mr. Philippe Krem. Να καλωσορίσουμε τον Φίλιππο ε, Ντεκρέμ που ήταν ε, πάρα πολύ δραστήριο τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Άμυνα και συγκεκριμένα όσον αφορά την ε, κοινή πολιτική Άμυνα. Σα υπενθυμίζω ότι ήδη διαδραματίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την προετοιμασία τη συζήτηση για το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στον αφορά την άμυνα τον Δεκέμβριο του 2010 στην Γάνδη. Γι' αυτό το λόγο και περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε τι θα βγει από το Συμβούλιο των Υπουργών όσον αφορά ε, τη συνάντηση κορυφής που θα γίνει φέτος τον Δεκέμβριο για την άμυνα. Και πιστεύω ότι και στην υποπιτροπή μα και στην ΑΦΕΡ ε, θα πρέπει να τάξουμε κάποιε προτεραιότητε, να τι προωθήσουμε και να προσθέσουμε όλα αυτά να τα περάσουμε το Συμβούλιο, να γίνει η Ευρωπαρασκευή, μια που είναι τόσο σημαντικό. Και ο κ. Ντονζόν θα σα πει τι προσδοκά το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο ε, εν ώψη αυτού του Συμβουλίου Κορυφή θα πρέπει να ε, προετοιμάσουμε τον δρόμο όσον αφορά για την ε, άμυνα και να υπάρχει έτσι συνεργασία για αυτό το ευθύτελευτική δίουλο που θα είναι το πλαίσιο για όλη αυτή τη διαδικασία και είναι ένα θέμα υψής σημασίας. Όλα αυτά ήδη περιέχονται στην σχετική μας ε, έκθεση η οποία πρότεινε και να συζητηθεί ενδελεχώς τον Οκτώβριο στην Επιτροπή μας. Επίσης διαπιστώσετε ότι τώρα προχωρούμε στη, στο θέμα της συνεργασίας. Ε, να δούμε τι θα γίνει με την ε, συνθήκη που έχουν έχει ολοκληρωθεί για τα θέματα της άμυνας που θα είναι τόσο σημαντικό για τόσε πολλές χώρε που θέλουν να προχωρήσουν στον τομέα αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει περισσότερο να χρησιμοποιήσουμε το συνασπισμό την ε, συνεργασία, να έχουμε τις ομάδες μάχης, να είναι πιο επιχειρησιακές, πιο λειτουργικές να είμαστε δημιουργικοί και από πλευρά τη βιομηχανία Γιατί θα πρέπει να έχουμε πιο ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Βέβαια είναι θέμα οικονομικό αυτό, αλλά αυτό μας κάνει αυτάρκης. Γιατί οπωσδήποτε και θα πρέπει να εξελίξουμε την υπάρχουσα ευρωπαϊκή πολιτική. Αλλιώς διακυβεύεται εδώ η εθνική κυριαρχία. Επίσης, έτσι, να δούμε πώς η συνεργασία μας επί τη βάση των όσων ε, θεσμικών πλαισίων έχουν συμφωνηθεί, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε με τη συγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό πλαίσιο. Έχουμε δεδομένο το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ασία, τη Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί τις πρώτες την ενέργεια, την τιμολογική της πολιτική για την ενέργεια σαν πολιτικό εργαλείο. Και στη συνέχεια έχουμε μια πολιτική αβέβαια Άρα και εμείς θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε προτεραιότητα τη σταθερότητα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Στο Βίλνιους είναι αυτή η διάσκεψη, την εθνικά κοινοβούλια και είδαμε πώς θα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Άμυνα πώς θα μπορέσουμε να πάμε σε κάποιο είδους υλοποίηση των όσων έχουμε αποφασίσει. Και βέβαια με τα 28 κοινά εθνικά κοινοβούλια συνεργαστήκαμε στενά σε σχέση με τα βασικά σημεία που πρέπει τώρα να προετοιμάσουμε εν ώψη της συνάντησης κορυφής του Δεκεμβρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο, επομένως, θα πρέπει να συνεργαστούμε με κάποιους ε, εξέχοντες υπουργούς όπως είστε εσείς για να δούμε πώς θα υπάρξει μια αυθεντική κατάσταση συνεργασίας. Να προσέξουμε τι θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Κορυφής, να μην έχουμε πενιχρά αποτελέσματα. Να φτάσουμε μόνο σε κάποιες και νέε περιεχομένου δηλώσει Να μπουν σε όλα αυτά τα θέματα, στην ουσία του, οι αρχηγοί κρατών και Και σα δίνουμε τώρα το λόγο. Ντονζό, σας ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε και πάλι, κύριε Υπουργέ. Είστε στο Κοινοβούλιο. Είσαστε τακτικό επισκέπτη συνεδριάσης μας και σα ευχαριστούμε και βεβαίως ε, ελπίζουμε ότι δεν έρχεστε μόνο μια που ε, βρίσκεστε εδώ κοντά μας γεωγραφικά, αλλά έρχεστε γιατί έχετε ενδιαφέρον για την ε, ΚΕΠΑ. Το Βέλγιο είναι ένας καλός μαθητής, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, και όσον αφορά το επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και όσον αφορά τη θεσμική πλευρά του θέματος, όσον αφορά την ΚΕΠΑ και τον ΝΑΤΟ. συμμετέχετε σε μια σειρά αποστολών και κάθε φορά σας έχει δοθεί ευκαιρία να δοκιμάσετε όλα τα θέματα που σας φαίνονται τα πιο επίμαχα σε σχέση με τη συνήθεια της Λισαβόνας, επίμαχα από συνταγματικής πλευράς και κρίσιμα για την ΚΕΠΑ και αν δεν κάνω λάθος είστε ο παλαιότερος των Υπουργών Άμυνα. Πριν από λίγε μέρε είχαμε στο Βίλνιου στην ε, Σύνοδο των Υπουργών Αμήνη, οπότε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να σα ακούσουμε και να διαπιστώσουμε ποιε είναι οι απόψει σα για τι πιο πρόσφατε εξελίξει. Και συγκεκριμένα ε, για τα όσα διακυβεύονται με τα οποία ασχολήθηκε το Συμβούλιο. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει απογοήτευση, δεν θα υπάρξει έλλειψη αισιοδοξία, γιατί νομίζουμε ότι θα πρέπει έκαστος να κάνει ό,τι μπορεί για να προετοιμαστεί σωστά αυτό το συνέδριο, αλλά τελικά αρχή κρατών και κυβερνήσεων θα δώσουν την επιθυμητή από όλους μας όθηση. Και επίσης θεωρώ ότι οι απόψεις του Ευρωκοινοβουλίου είναι ξεκάθαρες και σταθερές. Τα ξέρετε, τα Έχετε ακούσει, έχετε και την έκθεση της ε, κυρίας Κοπά. Είναι αυτή η γνωμοδότηση, αυτή η έκθεση η οποία πρόκειται να εγκριθεί το Νοέμβριο, δηλαδή που θα προηγηθεί του Συμβουλίου, οπότε και θέλουμε κάτι να γίνει. Ε, είχαμε και προηγούμενες εκθέσεις και τελικά ε, ήμασταν στο ίδιο μήκο κύματο αυτό το πρόσφατο παρελθόν. Να πούμε για την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Ε, πολλά Έχουμε το pooling and sharing και έχουμε και τη συμμετοχή σας σε μια σειρά επιχειρήσεων και επίσης και ε, υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα προτεραιότητα σε πολλά σημεία του κόσμου. Βεβαίως και στην άτυπη σύνοδο συζητήσατε για το Σαχέλ, για τη Συρία ε, και άλλα θέματα της Αφρικής. Όπως πάντα είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε με ενδιαφέρον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ Έλμαρ, αγαπητέ Αρνό. Με μεγάλη μου χαρά ήρθα σήμερα να σας συναντήσω και θυμάμαι την τελευταία συνάντηση. Που ήταν ενδιαφέρουσα για όλους ε, γιατί υπήρχαν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Γι' αυτό σας λέω ότι ήρθα εδώ, με ενδιαφέρον, με ικανοποίηση. Οπότε, χαίρομαι που υπάρχει ενδιαφέρον από την Επιτροπή Εξωτερικών του Κοινοβουλίου για τα θέματα της ε, άμυνας. Αυτό το θέμα που μας απασχολεί, που μας προβληματίζει, μια που το Δεκέμβριο θα γίνει η Ευρωπαϊκή Σύνοδος για την Άμυνα και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα προόδου για την ε, Ευρωπαϊκή Άμυνα. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας επομένως. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σαφές ότι θα πρέπει οι κυβερνήσεις να λάβουν κάποια μέτρα για την ε, άμυνα του Δεκέμβριου. και για το Βέλγιο. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να δούμε πώς θα καλύψουμε τις απόψεις των Ευρωπαίων και των εκπροσώπων τους. Ευχαριστώ για τη συμβολή σας. Με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα τις προτάσεις σας. Και επίσης ε, ευχαριστώ για την ενημερώση και άλλων συναδελφών υπουργών. Πριν πούμε στην ουσία, να σας πω κάτι πάρα πολύ βασικό για τη χώρα μου. Κάτι το οποίο πολλές φορές κινδυνεύει να αποτελέσει αντικείμενο σύγχυση. Εμείς είμαστε αναφαντών υπέρ της πρωτοβουλίας Φανεροπάε, ούτως ώστε το Δεκέμβριο στη Σύνοδο να γίνει ανοιχτή συζήτηση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα συζητηθεί το ίδιο σοβαρά όπως το περιβάλλον, όπως η επασχόληση, ε, το ίδιο θα και για την άμυνα. Άρα, έχουμε πολλούς λόγους να μην παραλείπουμε την άμυνα. Πρώτα-πρώτα έχουμε την πολιτική της λιτότητας. Θα πρέπει επίσης να αναπτύξουμε δυνατότητες τεχνολογικές, αλλά επίσης και τις ε, γεωστρατηγικές μεταβολές σε όλο τον κόσμο να τις λάβουμε υπόψη. Άρα, χρειάζεται συνεχής ε, προσπάθεια για να είμαστε θωρακισμένοι για να έχουμε πολιτική άμυνα. Θα πρέπει επομένω οι εργοί των κυβερνήσεων να στείλουν ένα μήνυμα αποφασιστικό το Δεκέμβριο. Μα δίνουν τη ευκαιρία τώρα να γραστητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τους ε, Ευρωπαίους για όλες τις ε, αλλαγές που γίνονται σε αναδειωμένες χώρες, σε πετροπαραγές χώρες ε, και όλα αυτά με τρόπο ανυφάλεια γιατί πολλές φορές έχουμε ε, τέτοιου είδους ζητήματα από αυτές τις χώρες γι' αυτό και χρειάζεται ένα ξεκάθαρο ζήτημα ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα μήνυμα το, οποίο θα είναι ολοκληρωμένο ούτως ώστε να μπορέσουμε και από τον πλευρά να μπορέσουμε να αυξήσουμε, να πλαισιώσουμε τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία δυνατοτήτων. Οπότε θέλουμε μία φορά το χρόνο να συζητάτε αυτό το ζήτημα στο Συμβούλιο. Δεν θέλουμε αυτό να γίνει μία φορά χωρίς επανάληψη, γιατί θα πρέπει ακριβώς αυτή η ιδέα, δηλαδή τα συμπεράσματα μια φορα χωρις επαναληψη γιατι θα πρεπει ακριβώ αυτη η ιδεα δηλαδη τα συμπερασματα μια συναντηση κορυφή, να συμβάλλουν ούτω ώστε να διαμορφώνονται προσπάθειες και τα θέματα αυτά έχουν να κάνουν με την ε, κυριαρχία, πολύ σημαντικό και γι' αυτό όλα αυτά θα αφορούν ένα μετασχηματισμό του πώς εμείς βλέπουμε την εθνική κυριαρχία. Αυτό άλλαξε τότε που υιοθετήσαμε το ευρώ, μια που είχαμε μια καινούργια οικονομική κοινή πολιτική. Έχουμε την κυρία Άστον, τις υπηρεσίες τις εξωτερικές και θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνουν όλα αυτά τα ζητήματα και έτσι να έχουμε τη, να προβληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσεχθεί τη βιομηχανία, αλλά προσοχή να μην κάνουμε λάθος ε, κίνηση. Θα πρέπει να προσέξουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν είναι τόσο εύκολο να τα πετύχουμε. Το Βέλγιο αυτό θέλει. Επίσης χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουμε κάποια τα αποτελέσματα τα οποία να είναι λειτουργικά deliverables λέμε στα αγγλικά και αυτό θα πρέπει να γίνει στη συνάντηση κορυφή. Είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε χρειάζεται για το Βέλγιο. Εάν δεν υπάρχουν αυτά αποτελέσματα, αυτό σημαίνει ένα μπούμεραν κατά των κυβερνήσεων. Αυτό θα δείξει μια παράλυση της πολιτικής ε, άμυνας. Οπότε Αυτά είναι πολύ σημαντικές ζητήματα που θα σας ε, τονίσω. Τώρα, για να δούμε τους τρεις βασικούς άξονες. Καταρχήν θα ήθελα να συμμιλήσω μαζί σας για την αποτελεσματικότητα της ΚΕΠΑ, όπως αναφέρθηκε από τον πρόεδρο Μπρόκ. Η επιχείρηση αυτή, αν και δεν στηρίζεται από μια από τη δημιουργία μιας εκστατείας επικοινωνίας θα πρέπει να βοηθήσει για να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι πολίτες κατά πόσο έχουμε μια αξιόπιστη, ε, έναν αξιόπιστο μηχανισμό αμήνης αυτός ο κόσμος δεν είναι τόσο ασφαλής όσο φαντάζονται οι, πολίτες, οι συμπολίτες μας. Οι σύγχρονες προκλήσεις είναι πιο απαιτητικές και θα μπορούσαν σοβαρά να επηρεάσουν την ασφάλεια όλων μας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν το γεγονός ότι η άμυνα έχει σημασία για μας. Δεν σημαίνει ότι δεν επειδή δεν κινητοποιείται ξένος στρατός στα σύνορά μας ότι δεν υπάρχουν απειλές για τη σταθερότητά μας και την ασφάλειά μας. Αυτή η αλλαγή είναι σημαντική για να μπορέσει η Ευρώπη σύντομα να αναπτύξει τις απαραίτητες δυνατότητες για να είναι σε θέση άμεσα και αποτελεσματικά και σε ανεξάρτητη βάση να αναπτύσσει στρατό που θα ενεργεί σε περιπτώσεις κρίσης στην επικράτειά της ή άλλο. Και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της ταχύτητας σε αυτό το πλαίσιο, σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων πριν από την ανάπτυξη στρατοβημάτων, καθώς και κατά τη διάρκεια αυτής. Αυτό είναι ο μόνος πιθανός τρόπος για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και τα συμφέροντά τους εντός και εκτός Ένωσης. Είναι όμως πεποίθησή μου ότι η Ευρώπη έχει να παίξει ακόμα πιο σπουδαίο ρόλο ε, σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο, εγκαθιστώντας τη σταθερότητα και την ειρήνη σε χώρες που έχουν πληγεί από συγκρούσεις. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με τους αντίστοιχους ε, διεθνείς οργανισμούς που είναι στρατηγικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς αυτό θα ήθελα να τονίσω επίσης τη σημασία της διατήρησης και της συντήρησης της στρατηγικού ηγετικού ρόλου με τους μη Ευρωπαίους εταίρους μας και τα πλονεκτήματα που έχει να κερδίσει η Ευρώπη ενεργώντας ως μια ενότητα σε αυτούς τους διαλόγους. Κυρίες και κύριοι, Πρόεδρε, συνάδελφοι, είναι αδύνατο να, θεωρήσουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στη θέση να προβεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως στη Λιβύη και στο Μαλί όντας λιγότερο εξαρτημένοι. Γιατί εμείς εστιάζουμε περισσότερο σε εκπαιδευτικέ αποστολέ, γιατί είναι ένα από τα ισχυρά μα σημεία και μπορούμε να προσφέρουμε προ αξία εδώ. Όμω γιατί οι ευρωπαϊκέ στρατιωτικέ μάχημε δυνάμει που είναι, εφ, εφ, ε, είναι σε θέση να αναπτυχθούν εντό 15 ημερών δεν έχουν κληθεί να συμμετέχουν σε στρατιωτικέ επιχειρήσει πέρα από το Μαλί, στην ευρωπαϊκή γειτονία η ευρωπαϊκή αντίδραση σε κρίση ήταν πάντοτε πολύ αργή και ακόμα και στο Μαλί ο χρόνος ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ανάπτυξης ήταν πολύ μακρύς. Αυτό είναι μια απλή και όχι πολύ ωραία αλήθεια. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά είχε ε, μπλεχτεί μέσα σε παγίδες ε, απόφασης, σε μακρές ε, τεχνικές συζητήσεις. Πρέπει να μπορέσουμε να αποφύγουμε και θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοια σενάρια στο μέλλον. Το πιο πολύτιμο μέσο, κυρίες και κύριοι, που έχουμε σε αυτό το θέμα είναι οι μάχημες μονάδες ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλωσορίζω το σχετικό έγγραφο που πρόσφατα εκδόθηκε και που διευκρινίζει τι, τι μπορεί να είναι μια τέτοια ομάδα, να είναι μια πραγματική μονάδα που δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να αναπτύξει γρήγορα, αποτελεσματικά και με ευελιξία στο σωστό μορφή που σημαίνει όχι απαραίτητο στο σύνολό τη αυτή την ομάδα, ώστε να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε είδο κρίση στην περιοχή τη το ε, Βέλγιο υποστηρίζει μία δυνατότητα προσαρμόσιμης ανάπτυξης, γιατί τα, στα θέματα αυτά θα πρέπει να είναι ε, εύκολα να πτυσσόμενα επιτόπου, να είναι ε, ευλίγιστα, ευέλικτα ε, και πολύ γρήγορα για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε αξιοπιστία ως Ένωση, ως αξιόπιστος εταίρος. Να θυμίσω δε ότι η ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα είναι η επιθυμία και τον ΗΠΑ, γιατί η Ουάσιγκτον ζητά πιο ισότιμη μοιρασιά του βάρους της ασφάλειας. Θα έλεγα λοιπόν να γίνει και μια εκδήλωση με αυτές τις ε, μάχημες μονάδες ε, στο μέλλον, με μεγάλη ορατότητα, μεγάλη δημοσιότητα και το ΝΑΤΟ διοργανώνει αντίστοιχε ε, συνεδριάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς, είναι, μια πολύτιμη, είναι πολύτιμο και είναι και απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο να εστιάσω στις αμυντικές μας δυνατότητες. Κυρίε και κύριοι, επί τόπου γνωρίζουμε ότι βραχυπρόθεσμα έχει ε, επιτευχθεί πρόοδος στο επίπεδο των περιφερειακών ε, συμπλεγμάτων. Ε, έχουμε προπολογισμού, έχουμε θεωτικό εξοπλισμό, στρατηγικό όραμα και εκτίμηση ε, για τις ε, απειλές. Αυτά είναι καταλητικοί παράγοντες ε, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και πρέπει να έχουμε τέτοια προσέγγιση σε περιφερειακή βάση. Πρέπει ωστόσο να προσέξουμε ώστε αυτές οι περιφερειακές δυνατότητες να μην αποτελέσουν τελικά τις δυνατότητες ολόκληρης ε, της ε, ε, Ένωσης ανά χώρα. Καλωσορίζουμε γι' αυτό την πρόταση της, Ιταλίας, να προχωρήσει στην ATC. Κατά τη γνώμη μου αυτός ο οργανισμός που έχει κρίσιμο ρόλο να πληρώσει είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, EDA. Θα πρέπει οι αρμοδιότητες της να αυξηθούν αντιστοίχως με την υποχρέωση φυσικά να δώσει αποτελέσματα. Γιατί αυτή η υπηρεσία θα παίξει ρόλο κλειδί στο συντονισμό, εποπτεία και καθοδήγηση της συνεργασίας ανάμεσα στα συμπλέγματα και στην ε, διάδραση ανάμεσα στα ίδια συμπλέγματα. Επιπλέον θα ήθελα να υπογραμμίσω το δυναμικό του άρθρου 44 της Συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπει στα κράτη-μέλη που επιθυμούν να προχωρήσουν γρηγορότερα να το πράξουν. Οι δυνατότητες που προσφέρει αυτό το θεσμικό όργανο θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφή του Δεκεμβρίου. Εν τέλει θα ήθελα να αναφέρω τη σημασία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην κοινή μα αυτή προσπάθεια. Έτσι όπως έχουμε το ευρύ και συμβατικό ε, θεσμικό τρίγωνο, δηλαδή Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν, θα πρέπει να έχουμε και ένα τρίγωνο που θα μας στηρίξει ώστε να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Ευρωπαϊκή Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αμήνης. Αλλά μπορεί να με ρωτήσετε αν η βάση της πρωτοβουλίας 2010 στη Γάνδη ε, ήταν ε, δεν έθεσε τη βάση ότι ε, η συνεργασία στην άμυνα είναι μια διαδικασία την οποία οθούν τα κράτη-μέλη. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά πρέπει αυτό να γίνεται από υπερκρατικά ε, υπερκρατικές διόδους γιατί έτσι κι αλλιώς οι σοβαρές ε, αποφάσεις περιεματικής πολιτικής θα πρέπει να γίνονται πλέον σε εθνικό επίπεδο. Και γι' αυτό και θέλω να καλωσορίσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα σημαντικό παίκτη στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία Άμυνας και ξέρω πως κάποια μέλη, κράτη-μέλη δεν το δέχονται αυτό εύκολα. Είμαστε σε μια καμπή κύριοι Ευρωβουλευτέ, και πρέπει να επιτύχουμε και να προοδεύσουμε. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει πολύ πιο θα πρέπει να γίνει πιο γρήγορα, αλλά και μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι μέχρι τώρα. Για να το πετύχουμε όλα αυτά έχουμε διάφορες επιλογές. Μπορούμε να έχουμε μια πολύ μακρά και φιλοσοφική συζήτηση για την ε, μεγάλη παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προσωρινώς να μείνουμε και να διατηρήσουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλεια του 2003 βάση και να σκεφτούμε ρεαλιστικά για τη γεωπολιτική θέση που θέλουμε να κατέχει η Ευρώπη σε παγκόσμιο πλαίσιο. Εγώ προσωπικά προτιμώ τη δεύτερη επιλογή. Επιπλέον, αυτό που είναι σημαντικό είναι να εντοπίσουμε τις στρατιωτικές δυνατότητες που απαιτούνται ώστε να διατηρήσουμε και να στηρίξουμε αυτή τη θέση. Όποια επιλογή και αν κάνουμε, χρειάζεται σαφής και σίγουρη εικόνα για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις δυνατότητες, την επικάλυψη και τα προγράμματα συνεργασίας. Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητές της ώστε να μπορέσει να ανακτήσει την κυριαρχία της σε στρατιωτικό επίπεδο. Ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναπτυχθούν κοινέ δυνατότητες στις στρατηγικές αεροπορικές μεταφορές, τον ανεφοδιασμό στον αέρα και στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Μισελ Μπαρνιέ, επίσης, ο αρμόδιος επίτροπος, επίσης καλεί για ανάπτυξη των δικών μας ε, μη επανδρομένων αεροσκαφών, των drones θα μπορέσουμε επίσης, θα πρέπει να, να απορροφήσουμε δυνάμεις από τον πολιτικό και από το στρατιωτικό κόσμο για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα θέλουμε λοιπόν συλλογική υπερεθνική οδό να ακολουθήσουμε στον τομέα της κυβερνοάμυνας ή είναι καλύτερη ο συντονισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη και πιο ρεαλιστικές βραχυπρόθεσμες λύσεις και πάλι. Το μεγάλο εμπόδιο σε αυτή την υπόθεση είναι και πάλι η κυριαρχία και το γεγονός ότι μια συλλογική προσέγγιση συχνά απαιτεί πολύ λεπτές πληροφορίες ε, ε, σε θέματα εθνικής ασφάλειας, οι οποία θα πρέπει να, γίνονται, ε, να κοινοποιούνται ανάμεσα στα κράτη. Τρίτο σημείο. Αμυντική βιομηχανία ή αμυντικές βιομηχανίες. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο για την ευρωπαϊκή μηχανή άμυνας που έχει κέρδη τζίρο 98 ε, δις ετησίως. Ε, είναι υπεύθυνη για 120.000 θέσεις απασχόλησης άμεσα και έμεσα για άλλες 400.000 ε, θέσεις απασχόλησης και είναι βασικός παίκτη όσον αφορά την ανάπτυξη και την γενοτομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία παίζει πολύ σημαντικό οικονομικό και τεχνολογικό ρόλο που δεν πρέπει να υποτιμάται στον τομέα της ευρωπαϊκής απασχόλησης και της διευκόλυσής μας να έχουμε απτά αποτελέσματα. Καλωσορίζω λοιπόν το γεγονός ότι η αμυντική βιομηχανία είναι κομμάτι κομμάτι του Horizon 2020 και επίσης θέλω να συγχαρώ την Κομισιόν για την ε, κίνησή της για αυτό το θέμα καθώς και για την έκθεση Ντάλερ. Τα πιεστικά ζητήματα που βρίσκονται επιτάπητος είναι τα εξής. περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς ε, αμυντικών εξοπλισμών και τη δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής βάσης ε, τεχνολογικής και βιομηχανικής άμυνας. Τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση από έξι μεγαλύτερες χώρες έχουν το 80% ε, της ε, αμυντικής βιομηχανίας και πολλές από τις εταιρείες ε, αυτές θεωρούνται από τις μεγάλες μεγαλύτερες μάλλον εταιρείε παγκοσμίω. Υπάρχει όμως τεράστιο βιομηχανικό δυναμικό εκτός αυτών των έξι χωρών. Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν στο full δυναμικό τους γιατί γιατί αυτή τη στιγμή εφαρμόζουν, μάλλον εκτελούν τις παραγγελίες που λάβαν πριν από 10-15 χρόνια. Συχνά προσφέρουν δε την εμπειρογνωμοσύνη τους σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η παρατήρηση μας φέρνει άμεσα στην συζήτηση ε, όσον αφορά τα, τις αντισταθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητα των αμυντικών μας βιομηχανιών. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, εξάλλου, αυτή τη στιγμή ε, μπορούν να φτιάξουν ε, πρωταθλητές εθνικής άμυνας και να γίνουν εμπειρογνώμονες. Σύντομα θα είναι αδύνατον θα είναι αδύνατον οι δικές μας επιχειρήσεις να ακολουθήσουν αυτήν την πορεία. Ε, πρέπει δε να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε άμεσες και ε, έμεσες αντισταθμίσεις. Οι τελευταίες είναι πολύ βλαβερές τα ευρωπαϊκά μας προγράμματα. Δεν μπορούμε να εξάγουμε εξαιρετικό εξοπλισμό που εξαρτάται από την υποχρεωτική αγορά άσχετων αγαθών όπως ε, τάπητες ή ελαστικά. Ωστόσο, με την, την, την, μεταφορά τεχνολογίας μπορούμε να συμβάλλουμε στην, στον κατακαιρματισμό της, βιομηχανία, της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Κυρίε και κύριοι, επιπλέον τα κράτη-μέλη ε, ε, τα έχουν πάει καλά. Έχουν μεταγράψει την οδηγία περί αμυντικών προμηθειών το 2009 σε εθνική νομοθεσία. Αλλά τι γίνεται με τις πρακτικές επιπτώσεις της. Για να έχουμε σαφή εικόνα για τις εξελίξεις εκεί, θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τους όρους των συμβάσεων, τα αγαθά που παράγονται σε, σύνδεση με εκείνη την ε, πρωτοβουλία του 2009 θα πρέπει να δημοσιεύονται όπως ε, στην ε, καθημερινή ηλεκτρονική βάση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν για τους ε, μειοδοτικούς διαγωνισμούς είτε στο πίνακα επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αμήνης. Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς ε, της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν γίνεται κάτι τέτοιο συστηματικά. Η αμυντική βιομηχανία πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστική και πιο ανοιχτή για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί όλα τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. Η πρόκληση είναι ότι πολλές χώρες δεν ε, ερμηνεύουν την πραγματική έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης Υπερλειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν τον τρόπο και διατηρούν αμυντικά προϊόντα εκτός της κοινή πρακτικής της εσωτερικής ε, αγοράς. Χρειάζεται να βρεθεί μια λύση για αυτό το θέμα. Τέλος, καλύτερη εικόνα για την ευρωπαϊκή αγορά αμυντικών προϊόντων έτσι ώστε οι πολιτικοί φορείς αλλά και οι φορείς του τομέα να έχουν καλύτερη εικόνα για τις εξελίξεις στον τομέα. Αυτό ακόμα σήμερα δεν ισχύει. Πιθανές λύσεις τώρα θα ήταν να τονίσουμε τα δυνητικά μεγάλα ε, πλονεκτήματα ε, της ε, προμήθειας ετοιμοπαράδοτων προϊόντων ως ένα ενδιαφέροντα τομέα για να αποφευθούν οι καθυστερήσεις τα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα θα, πρέπει, ε, θα εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο εναρμόνισης και θα οδηγήσουν ε, στην χρήση από περισσότερα έθνη του ίδιου εξοπλισμού και άρα θα αυξηθεί και η διαλειτουργικότητα. Γι' αυτό και συγχαίρω την ε, πρωτοβουλία περί αποτελεσματικών προμηθειών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αμήνης. Και τώρα κυρίες και Αγαπητοί φίλοι, να φτάσουμε στα συμπεράσματα, μια που πάρα πολύ λίγο χρόνο πριν την συνάντηση κορυφή του Δεκεμβρίου. Εν τω μεταξύ, όλο ο κόσμο μπόρεσε να σχολιάσει, να αναλύσει τα δύο βασικά κείμενα, δηλαδή την έκθεση τη ε, υπάτη εκπροσώπηση κυρία Άστον και την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ονομάζεται ω μια ε, πιο αποτελεσματική ε, πολιτική για την άμυνα και την ασφάλεια. Επίσης έχουμε διάφορες άλλες χώρες οι οποίες έχουν ε, συντάξει πάρα πολλά άλλα ε, έγγραφα και κάθε φορά υπάρχουν και ενδιαφέρουσες ιδέες. Έχουμε επίσης την σύνοδο του, του Σεπτεμβρίου κατόπιν τον Κίμνικ των Υπουργών Εξωτερικών και έτσι μπορέσαμε να μάθουμε τις απόψεις τους. Τώρα πέραν αυτού νομίζω ότι η πάτη εκπρόσωπος θα πρέπει τώρα όσο αυτό είναι δυνατόν να βελτιώσει ακόμα και να ολοκληρώσει την εκθεσή της και να εμείνει στις τρία θέματα τα οποία θα σας εξηγήσω. Πρώτα-πρώτα την ενίσχυση της στρατηγικής οπτικής και οράματος, την αναζήτηση περισσότερων συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και το πώς θα φτιάξει όσο είναι πιο συγκεκριμένο χάρτη πορείας για τους ε, στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς οι κυβερνήσεις του Βελγίου θα προσέξει τα θέματα γιατί το ενδιαφέρον αυτής της έκθεσης και των συμπερασμάτων θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα να σας πω κάποιες γενικές σχέσεις ενίδη συμπερασμάτων, κάτι το οποίο θα μας ε, δώσει την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε τις εργασίες ε, του Συμβουλίου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Πρώτα-πρώτα, η τωρινή ε, προβληματική είναι πρώτα-πρώτα ε, πολιτικού χαρακτήρα περισσότερο παρά στρατιωτική, στρατιωτικού χαρακτήρα. Γιατί η πολιτική δίνει την όθηση στους στρατιωτικούς και τα μέσα ούτως ώστε να μπορέσουν να κινηθούν στην παγκόσμια σκηνή, γιατί χωρίς να υπήρχε πολιτική όθηση τίποτα σχεδόν δεν μπορούσε να γίνει. Επομένως, από τις κυβερνήσεις να λάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν στην άμυνα ε, τον, τον, ρόλο που τις ε, αρμόζει. Η δε συνάντηση του Δεκεμβρίου ακριβώς προσφέρει στους αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων μια μοναδική ευκαιρία για να μπορέσουν να εντάξουν την άμυνα ή στην υπόθεση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και αν δεν, όπως ε, όλοι ε, από ό,τι φαίνεται το δέχονται, ε, έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινές αξίες και δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε κι άλλο στα θέματα συνεργασίας και ελληνικής όσον αφορά την, την άμυνα. Χρειάζεται και μέσα σε μια τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινών Αξιών εμείς δεν θα πρέπει να όλοι στένουμε σε, σε, ατομισμούς και εθνικισμούς γιατί θα πρέπει ε, αυτό που έχει σημασία να έχουμε μια κοινή άμυνα. Μια επίθεση κατά ενός θα πρέπει να θεωρηθεί επίθεση κατά όλων. Και αυτό είναι πριν ένας ε, κανόνας ο οποίος ε, ισχύει 100%. Επίσης έχουμε την συντριπτική πλειοψηφία των ειδικών από πλευράς άμυνας που συμφωνούν ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα σήμερα δεν είναι δυνατόν μόνη της να να, να, να, να υποστεί μια επίθεση μεγάλου βεληνικούς ε, απομονωμένη. Δεν μπορεί να κάνει κάποια επιχείρηση ε, σε κάποιο θέατρο επιχειρήσεων μακριά από την Ευρώπη. Χρειάζεται επομένω ε, μια συνεργασία, ένα συντονισμό που επιβάλλονται για λόγου τεχνολογικού και οικονομικού. Ο πιο ισχυρό μα σύμμαχο, δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, επιθυμεί οπωσδήποτε να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα ως Ευρώπη. Χρειάζεται επομένω μια κατανομή του σχετικού άχθους για την άμυνα, ε, μια κατανομή πιο δίκαιη και αυτό δεν μπορεί πλέον να έχει ως, μόνο επιχείρημα κατανομής στην στρατιωτική ενωνετρότητα τον είπα. Εάν θέλουν οι Ευρωπαίοι να είναι αξιόπιστοι σύμμαχοι, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες για την άμυνα. Και για να μπορέσουμε να πάμε σωστή κατεύθυνση, οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε πιο αποφασιστική ε, ηγεσία ε, που να προβάλλεται περισσότερο γιατί χρειάζεται λέει, το Βέλγιο επίσης μεγαλύτερη συνεργασία ε, μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων στην Ευρώπη, δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επομένω να γίνεται κάτι τέτοιο γιατί έτσι δεν τίθεται να αμφιβόλω οι άλλες συνεργασίες συνεργασίες με τις μικρότερες χώρες. Όπως γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ ε, βασική συνεργασία με τις κάτω χώρες και το Λουξεμβούργο. Γνωρίζετε πόσο το, το Βέλγιο αποδίδει σημασία σε αυτή τη συνεργασία. Όσον αφορά τώρα την περιφερειακή συνεργασία, έχουμε την ομάδα του Βίσεγκρατ και έχουμε τις ε, χώρε της Σκανδιναβίας και, αυτές, αυτοί οι φορείς, αυτές οι πλατφόρμες υπόσχονται πολλά και γι' αυτό το λόγο το Βέλγιο ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε, ότι βοηθά τη συνεργασία μεταξύ των τριών μεγάλων. Και αυτό θα διευκολύνει το έργο των μεγάλων. Και αυτοί μπορούν επίση έτσι να προσφυλωθούν περισσότερο στα σχέδια και στα όσα έχουν αποφασίσει να γίνουν. Και γι' αυτό και εμένα ότι θα πρέπει να έχουμε τέτοιο προγραμματισμό ε, μεταξύ του, των όσων θα κάνουν οι Ευρωπαίοι το, τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιες κοινέ αποφάσεις, να έχουμε συμβατά συστήματα και α, βεβαίως η ωφέλεια εδώ πέρα είναι αυτονόητη. Για να κλείσω τώρα. Αυτό που θα να σας πω είναι να σας πω ότι χρειάζεται ε, να αναδεχθούμε και να συμφωνήσουμε ακόμα περισσότερο όσον αφορά με τα θέματα της εθνικής κυριαρχίας είναι κάτι που είναι τα Άγια των Αγίων για, για πολλούς αυτή η έννοια. Όμως δεν έχει απόλυτο χαρακτήρα αυτός, αυτή η εθνική κυριαρχία σε ε, κανένα τομέα. Γιατί κανένα κράτος δεν μπορεί να ζει ε, απομονωμένο ε, και να θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητο το τι κάνει, την πολιτική ακολουθία 100%. Γι' αυτό και λόγω της, του πρώτης παγκοσμιοποίησης οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν πιο εντατική συνεργασία σε όλους τους τομείς, στην οικονομία, στο περιβάλλον, αλλά και στην άμυνα, για να αντιμετωπίσουν τις εξωτερικές πιέσεις. Η αυθεντική, η αυθεντική είναι αυτή την οποία την μοιραζόμαστε. Κυρίε και κύριοι, με αυτό το πνεύμα το Βέλγιο και η Βελγική κυβέρνηση θα κατέβουν στην ε, διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου. Η χώρα μας θα δεχθεί όλα όσα βοηθούν ούτω ώστε να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ε, πιο ολοκληρωμένη, πιο ισχυρή. όσον αφορά την άμυνα. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαρίστω να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσει έχετε πάνω στην εισήγησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκάθαρα όλα. Ήδη έχουμε ε, προτρέξει των εργασιών του Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ που αγγίξατε όλα τα θέματα. Ήταν μια comprehensive approach, όπως θα μας έλεγε η αγαπημένη μας ύπατη εκπρόσωπος. Ε, ε όντως αγγίξατε όλα τα θέματα και φαντάζομαι θα προκαλέσει αυτό ερωτήσεις και σχόλια. Και ο αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος μας... Ο κύριος Σοφοκλέος θέλει να πάρει το λόγο. Καταρχάς με την σειρά μου πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Υπουργό για την ολοκληρωμένη του παρέμβαση. Θα περιοριστώ μόνο σε μια ενότητα στην αμυντική βιομηχανία την οποία θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε δύο πράγματα στο πρώτο το οποίο έχει ακουστεί ότι αποτελεί μια οικονομική ισχυρή δύναμη και μόνο από τα έσοδα μιλούν, μιλά από μόνη της 98 περίπου δις. Η δεύτερη θέση και που πρέπει να συμφωνήσουμε ότι και εδώ όμως υπάρχει μια διάσπαση, ας μου επιτραπεί η έκφραση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Δηλαδή έχουμε έξι ισχυρέ χώρες που καλύπτουν περίπου το 80% της αμυντικής βιομηχανίας. Και αφού ο στόχος μας είναι να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, η αμυντική βιομηχανία πιο ανταγωνιστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Υπάρχει, πιστεύετε, ένα σχέδιο, συγκεκριμένο σχέδιο, που μπορεί να ενώσει, θα έλεγα, σε αυτόν τον τομέα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση πρώτον της κοινή έρευνα για τα εξοπλιστικά συστήματα για να υπάρξει λιγότερο κόστος. Δεύτερον, να μην υπάρχει επικάλυψη από μία χώρα σε άλλη. Και τρίτον, πολύ σημαντικό, αν μπορεί να υπάρξει ένας ενιαίος αμυντικός σχεδιασμός ε, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από σήμερα. Διότι όλοι συμφωνούμε ότι κάποτε πρέπει να υπάρξει αλλά πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και να δώσουμε αυτή την, σε αυτή την έννοια περιεχόμενο απέναντι στις ΗΠΑ, Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία νομίζω, μόνο ενωμένε οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλώ πάντοτε για τα εξοπλιστικά συστήματα. Βλέπετε να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, τέτοια προοπτική, όχι επιθυμία, δυνατότητα προοπτική πρακτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως για τη φιλοδοξία και τη δέσμευση που επιδεικνύεται πριν από την Σύνοδο του Δεκεμβρίου και να επαναλάβω αυτά που είπατε για την κυριαρχία. Μιλάμε για δύο σκέλη. Καταρχάς, κυριαρχία σημαίνει να μπορεί να λάβει κανείς μια απόφαση, αλλά και να την εφαρμόσει μόνο του. Και στο βαθμό που δεν είμαστε σε θέση να τα εφαρμόσουμε αυτά μόνοι μας, ε, μιλάμε για shared sovereignty πλέον, ε, κοινή τέτοια επικυριαρχία. Και γι' αυτό λοιπόν Έχετε δίκιο. Σα ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σύμφωνο απολύτω και συμφωνώ επίση ότι πρέπει να επιταχύνουμε τι αποφάσει λήψη, ε, τι ε, διαδικασίε λήψη απόφαση. Ερωτήσει που έχω να σα απευθύνω συγκεκριμένα. Θα ήσασταν υπέρ για την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων που θα λεφτούν το Δεκέμβριο να γίνει πιο επίσημη η διαμόρφωση του Υπουργείου, των Υπουργών ε, Άμυνας, όχι μόνο για να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις δηλαδή και όχι μόνο για να συνοδευτούν αυτές οι αποφάσεις. Και πιστεύετε ότι μία απόφαση θα πρέπει να είναι μία, να συμφωνήσουμε ε, επί μίας αναθεώρησης ε, της άμυνας, δηλαδή να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και τι χρειαζόμαστε επιπλέον. Τρίτη ερώτηση αν σωστά κατάλαβα, είσαστε υπέρ της ενίσχυσης του, α, της α, ε, λειτουργίας συντονισμού της EDA, της υπηρεσίας ε, α, Σε ό,τι αφορά το σχέδιο άμυνας, ε, σε ό,τι αφορά τη, τα θέματα ζήτησης, θα μπορούσατε να το επιβεβαιώσετε αυτό ότι θέλετε να έχει πιο έντονο συντονιστικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο η EDA και σε ό,τι αφορά το στάτους της ε, EDA για το 2014 που θα πρέπει να αποφασίσουμε εκ νέου. σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το προσωπικό της EDA θα μπορούσε να πληρωθεί στο μέλλον από τον προπολογισμό της Επιτροπής. Μία άλλη ερώτηση για την εσωτερική αγορά σε ό,τι αφορά τα αμυντικά προϊόντα έχουμε αυτό το άρθρο 346 με το οποίο πατάνε φρένη τα κρατημέλη και μιλάνε για εθνικά σημαντικά συμφέροντα και αποσύρονται από την ενιαία αγορά. Θα υποστηρίζατε μια πιο αυστηρή διαμόρφωση από πλευράς της Κομισιόν των σχετικών προτύπων. Σε ποιους τομείς θα ήσασταν υπέρ μιας μελλοντικής ε, δομημένης μόνιμης συνεργασίας. Θα μπορούσατε να πείτε ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή ένα τέτοιο εργαλείο και τέλος ότι αφορά τυποποίηση και πιστοποίηση. Φαίνεται ότι δεν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδο στο ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό της τυποποίησης δεν μπορούσε να βοηθήσει η Γαλλία και η Γερμανία σε ό,τι αφορά το refueling LTR. Θεωρείτε ότι μπορεί να κάνουμε κάτι παραπάνω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Merci. Madame Coppa. Εκτός μικροφώνου. Thank you. Uh, Σας ευχαριστώ για πολλούς ε, εξημών. Uh, η Σύνοδος του Δεκεμβρίου είναι κάτι το οποίο περιμένουμε ε, με ανυπομονησία, γιατί το είχαμε συζητήσει ήδη και πέρσι το θέμα αυτό. Λοιπόν, επειδή πιο πολλοί από εμά θεωρούμε ότι τα θέματα άμυνας ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να θέσουμε στην προεκλογική εκστρατεία, θεωρώ ότι σημαντικό θα ήταν να γίνει μια ένα follow-up στην Σύνοδο του Δεκεμβρίου δεν θα έπρεπε να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός και θα ήταν σημαντικό και ενδιαφέρον από πολλές ε, απόψεις να υπάρχει ένας οδικός χάρτης για τις επερχόμενες δράσεις, να υπάρχουν ορόσημα, benchmarks και να συμφωνήσουμε σε κάποια επόμενη ημερομηνία. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε θέματα άμυνας σε μια βάση ad hoc. Ξέρουμε ότι σε εποχές οικονομικής κρίσης Πολλά από τα κράτη-μέλη και πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άλλωστε δεν πιστεύουν ότι θέματα άμυνας θα έπρεπε να είναι στην ατζέντα. Αυτό είναι κάτι απολύτως εσφαλμένο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πολιτών μας. Είναι κάτι το οποίο απαραίτητο πρέπει να τεθεί επιτάπητος. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να ακούσω την άποψη του Βαλγίου επ' αυτών και να διασφαλίσω ότι αυτά που έθεσε ως ερωτήματα ο συνάδελφος Γκάλερ για το ρόλο της ΙΝΤΑ θα απαντηθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της EDA σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι ικανοποιημένα ιδιαίτερως όταν δίδεται με το ενδεχόμενο Ανάθεση άλλε εντολής στην EDA σε ό,τι αφορά δηλαδή, την ενίσχυση του ρόλου τη. Πείτε μα και εσεί όμω τη γνώμη σας. Ευχαριστώ. Κρίστοφ Λίζεκ που μόλις ήρθε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, εκτιμώ ιδιαίτερο το γεγονό ότι μιλάτε εδώ και πολλά χρόνια για τα θέματα αυτά. Νομίζω πριν από κάποια χρόνια στο Χάλεφαξ είχατε αναφέρει τα ίδια πράγματα. Είσαστε συνεπείς λοιπόν και συνεχίζετε να τα επαναλαμβάνετε αυτά με συνέπεια. Πολλοί συνάδελφοι έχουν θέσει ήδη κάποια ερωτήματα τα οποία με απασχολούσαν και εμά. Και εσεί έχετε ήδη απαντήσει σε δύο ερωτήματα που είχα προετοιμάσει. Ένα σχόλιο, μία ερώτηση λοιπόν έχω να κάνω. Το σχόλιο για το pooling and sharing, το οποίο το αναφέρω και στην έκθεση μου πριν από δύο χρόνια, στην έκθεση που ολοκλήρωσα πριν από δύο χρόνια για τι συνέπειε τη οικονομική κρίση. Ασφαλώς αυτό το pooling and sharing έχει ω αποτέλεσμα κάποια εξοικονόμηση, αλλά δεν αρκεί αυτό γιατί οι εμπειρογνώμονε υπολογίζουν ότι τα project που έχουμε τώρα ίσω αποφέρουν 300 εκατομμύρια αποταμιεύσει Οι δε περικοπέ, είναι ε, εκατονταπλάσιε στα κράτη-μέλη. Άρα δεν αρκεί αυτό. Η ενίσχυση της βιομηχανίας είναι ε, μια μεγάλη πρόκληση και θα μας πάρει πολλά χρόνια, γιατί για παράδειγμα κρατημέλη σίγουρα θα προστατεύουν τις θέσεις εργασίας ε, στις ε, στρατιωτικές τους εταιρείε. Τώρα, το ερώτημα είναι... Είπατε ότι δεν έχουμε εχθρούς πρώτων συνόρων μας. Αληθεύει αυτό. Από την άλλη όμως, Έχουμε τις ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας. Θεωρητική νομίζω, ελπίζω, είναι η υποτιθέμενη επίθεση στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οικονομική και πολιτική πίεση αντιμετωπίζουμε επίσης από τη Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Άρα, ερωτώ, μήπως θα έπρεπε να συνεργαστούμε στενότερα και στον τομέα της άμυνας με τις χώρες Ανατολικής Γειτονίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φανόρντον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Υπουργέ Αμυνα για τα σχόλιά σας. Συναρπαστικά. Κάποιες ερωτήσεις έχω να κάνω. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επωφελούταν από μια, ένα προπολογισμό ξεχωριστό για την άμυνα δικό τη Θα υποφελούνταν επίσης από μια πιο ενοποιημένη δομή εντολών και διαχείρισης. Και πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Ευχαριστώ, κυρία Κόμες. Κύριε Υπουργέ, Συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι δεν αρκεί το pooling and sharing. Να σας ρωτήσω κατά πόσον θεωρείτε ότι υπάρχει όρεξη και θα εκδηλωθεί αυτή στην σύνοδο του Δεκεμβρίου για να αναφερθεί το σύστημα χρηματοδότησης της ΚΕΠΑ. Το παρόν σύστημα και το κόστος του είναι επιβλαβές σε ό,τι αφορά την δημιουργία δυνάμεων στα πλαίσια των επιχειρήσεων και πά. Θα μπορούσαμε σε ό,τι αφορά τη δημιουργία, για παράδειγμα, και την αποστολή στρατευμάτων, ε, δεν υπάρχουν δυνατότητες, γιατί μας ε, έχει ε, βάλει σε ασφακτικό κλειό η κρίση και η λιτότητα. Άρα, το να υπάρχει διαφορετικό burden sharing ε, κατανομή του βάρους το να επιτρέψουμε ουσιαστικά στα κρατημέλη να έχουν ε, στρατεύματα τα οποία να μπορούν να αναπτύξουν θα δημιουργούσε μια διαφορετική κατάσταση σε ό,τι αφορά και τις ε, επιχειρήσεις της ΚΕΠΑ, όπως για παράδειγμα στο Μάλι. έχει να κάνει και με τη Συρία. Αναρωτιέμαι, το έχουν συζητήσει αυτό οι Υπουργοί Άμυνας σε χώρες, για παράδειγμα, όπου αντιμετωπίζουμε οικονομική κρίση, όπως ε, στη δική μου τη χώρα, την Πορτογαλία. Είναι πραγματικά εξοργιστικό ότι η Τρόικα δεν υπολογίζει τις συνέπειες ό,τι αφορά την ανάπτυξη τέτοιου δυναμικού για περιπτώσεις ε, τέτοιες. Δεν έχουμε, για παράδειγμα, χρήματα για να βάλουμε καύσιμα στα υποβρυχιά μας. Για να βγουν στα χωρικά μας ύδατα, όχι για να κάνουν τίποτα το μεγαλόπνο, αλλά για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και εμεί δεν έχουμε χρήματα για να βάλουμε καύσιμα σε αυτά τα υποβρύχια. Και αυτό νομίζω ότι εξηγεί εν μέρη γιατί έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει η χώρα μου. Για το θέμα α, της θαλάσσης πολιτικής σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της διόρυγας του Παναμά, για παράδειγμα. Αυτό έχει τεράστιες ευκαιρίες, αλλά ναι, έχει και τεράστιους κινδύνους σε ό,τι αφορά τις εγκληματικές δραστηριότητες στον Ατλαντικό. εξετάζεται το πώς διαμορφώνονται τα σύνορα και πώς ε, αλληλοεπικαλύπτονται τα σύνορα μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας. Ε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια, χρειαζόμαστε μια κοινή εκτοφυλακή. Για παράδειγμα, στη, χώρα μου, στη χώρα μου ε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίπλοκια. Ε, σε άλλο τομέα μπορεί να παρέμβει η ακτοφυλακή, σε άλλο η χωροφυλακή, η αστυνομία. Αυτό δεν έχει αποτελέσματα ούτε για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ούτε για την εθνική ασφάλεια. Και τέλος, να σας ρωτήσω, η επιχείρηση για τη Λιβύη, την οποία το Κοινοβούλιο ζητούσε επί σειρά μηνών για την ε, στρατιωτική επιχείρηση και μετά η επιχείρηση όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στα σύνορα, η οποία τώρα μόλις ξεκινά, αλλά για την ασφάλεια την περιφερειακή της Λιβύης και τη δική μας την ασφάλεια άλλωστε. Για την εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων Και τώρα, η Λιβύη μας το έχει ζητήσει αυτό επανειλημμένα και τίποτα δεν έχει συμβεί. Και τώρα το πράγμα έφτασε στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ θα, το, θα ανταποκριθεί. Αυτό τι σημαίνει ότι πάλι εμείς θα το κάνουμε, μιας και εμείς είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ πιο πολύ. Γιατί δεν το έχουμε κάνει λοιπόν αυτό, λείπει πολιτική βούληση. Και αυτό με τι σχετίζεται, τα κράτη-μέλη θέλουν να συνεχίσουν ε, με την υφιστάμενη κατάσταση χωρίς να εντρώνουν αυτοί του και χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό είναι πολύ επιζήμιο για τη δική μας ασφάλεια. Πείτε μας λοιπόν πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Πού βρίσκεται η συζήτηση. Στο Συμβούλιο των Υπουργών Αμήνη. Oui, monsieur. Ο κ. Λανσπέργης και μετά θα δώσω το λόγο στον κ. Ντεκρέμ για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομο σχόλιο. Μετά από αυτά που είπε και ο προηγούμενος συνάδελφός. Φυσικά πρέπει να δυσφαλίσουμε ότι δεν έχουμε εχθρούς προς το σύνορων μας. δεν έχουμε εχθρούς, αλλά έχουμε ανθρώπους που μας θεωρούν εμάς εχθρούς. Αυτό νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ce fut effectivement bref. Ήταν πραγματικά σύντομο και σαφή. Ο κύριο Υπουργό έχει το λόγο για να απαντήσει. Answer in the opposite way, and I will start with the remark that was made by President Landsbergis. Um, για να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κ. Λανσπέργης, ε, καταλαβαίνουμε τι αντιμετωπίζουμε. Σε αυτή τη φάση το Βέλγιο συμμετέχει στην, ε, σε ένα πρόγραμμα ελέγχου του ε, Βαλτικής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι εννοείται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας απασχολεί ιδιαίτερως. Αν αναπτύξουμε ένα όραμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το σύντομο μήνυμα το οποίο μεταφέρατε. Πολλοί συνάδελφοι ρώτησαν ποιος είναι ο σκοπός, ο στόχος της Συνόδου του Δεκεμβρίου. Καταρχάς, να σας πω ότι οι Υπουργοί Αμήνης δεν θα συμμετάσχουν στην συνάντηση. Ίσως ο Υπουργός Εξωτερικών να συμμετάσχει στην συνάντηση και αν ναι, συμμετάσχουν οι Υπουργοί Οικονομικών, ε, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσέξουμε γιατί πολλοί συνάδελφοι σε εθνικό επίπεδο όταν μιλούν και αθρίζουν τα ποσά που έχουμε και που δαπανούνται για την άμυνα διαπιστώνουν ότι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι πηγαίνει ακόμα στην άμυνα. Να το έχουμε υπόψη μας ότι δεν έχουμε μόνο φίλους αλλά και εχθρούς στην σύνοδο του Δεκεμβρίου. Και θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιο θα πρέπει να είναι ο στόχο τη Συνόδου του Δεκεμβρίου. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ, να κοιτάξουμε το επιχειρησιακό σκέλο, όχι τόσο πολύ να εστιάσουμε στην ιστορία, αλλά να κοιτάξουμε και τα διδάγματα τη ιστορία. Το είπε αυτό ο κ. Λαντσμπέργκη και άλλοι συνάδελφοι. Αλλά και το τι μα διδάσκουν τα πιο πρόσφατα γεγονότα. Να δώσουμε μια απάντηση στο γεγονό, ε, στο πού είναι οι ελλείψεις μας, πού είναι τα κενά μας. Το είδαμε αυτό και σε πρόσφατες επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετείχαν και κάποιες χώρες εδώ πέρα. Τι μας ε, έλειπε, τι, ποιο ήταν το πρόβλημα στο Μάλι που ξεκίνησε η Γαλλία και συνέχισαν οι υπόλοιπες χώρες. Χρειαζόμαστε καύσιμα, χρειαζόμαστε ανταλλαγές μέσω δορυφόρων, χρειαζόμαστε μη επανδρομένα τέτοια αεροσκάφη. Αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα της δουλειάς που έχουμε να κάνουμε το Δεκέμβριο. Μια ρεαλιστική λοιπόν προσέγγιση. Δεν πρόκειται για ένα πρώτο τμήμα μιας ευρωπαϊκής άμυνας, όχι. Αλλά θα πρέπει να, το, να δούμε τι χρειάζομαστε. Επίσης να δούμε τι θέλουμε να σημαίνει στους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς. Είναι, μπορούμε να αναπτύξουμε τις δυνάμεις μας. Η πρόταση που έκανα είναι τα, ε, τα που συμμετέχουν στις μάχημες ομάδες να έχουν κάποιες δυνατότητες και μετά να αποφασίζουν ποιο τμήμα θα μπορεί να αναπτύσσεται των μάχημων ομάδων. Επίσης κάποιοι αναφέρθηκαν στο τι συνέβη στη Λιβύη. Είχα μία συμφωνία Καταρχάς θα πρέπει να γίνει το στρατιωτικό σκέλος ε, του επιχειρήματος υπό την γύβα των Ηνωμένων Εθνών με το καθεστώς Καντάφη και το καθεξής. Υπήρχε λοιπόν αυτή η στρατιωτική επιχείρηση 100% εστέφθη με επιτυχία. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία λήψης απόφασης και υπήρχε και ένα θέμα της αλληλεγγύης εντός του ΝΑΤΟ. Δεν είναι καλό το γεγονός ότι μόνο εννέα κράτη-μέλη συμμετείχαν. Τι έγινε όμως μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να κάνουν τη δική τους δουλειά για την ανάπτυξη δυναμικού στην κοινωνία των πολιτών, στον κοινωνικού ιστού. Αυτό δεν λειτουργήσε. Μπορούμε να το αναφέρουμε ότι το κρατάμε ως μάθημα, αλλά αυτό δεν θα συζητηθεί το Δεκέμβριο απαραίτητα. Σε ό,τι αφορά, κυρία Γκόμες, αυτά που έχει και χρειάζεται η πορτογαλική κυβέρνηση. Δεν είναι δικός μου ρόλος να σχολιάσω αυτά. Να επανέλθω σε ένα άλλο ζήτημα όμω. Είναι πραγματικά κάτι που δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ότι μπορούμε να αναπτύξουμε ένα όραμα χωρίς τον σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να παίξει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του οράματος. Αυτές τις τρεις χώρες θα πρέπει να συμμετάσχουν επίσης ορούς και θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να αντιδραματίσουν. Πρόκειται για μια ανάληψη ευθύνης για ε, ανάπτυξη του ευρύτερου σχεδίου στο οποίο θα ενταχθούμε. Άρα θα πρέπει να είναι λειτουργικό όλο το πρόγραμμα της Συνόδου και θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε να κάνουν αυτές οι μάχημες ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εννοώ ότι θα πρέπει να μάχονται, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείουμε ότι υπό τους όρους που θα ορίσει η Ευρώπη, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, ένα τμήμα των μάχημων ομάδων αυτών θα μπορέσουν να αναπτυχθούν σε μια ενδεχόμενη μελλοντική αποστολή. Και έτσι νομίζω ότι απάντησα και στο ερώτημα που έθεσε ο συνάδελφος Φανόρντεν. Όχι, δεν σας απάντησα. Α, για τον προπολογισμό. Τα κονδύλια. Κοιτάξτε. Βλέπω ότι όλα τα κρατημέλη αντιμετωπίζουν την τεράστια πρόκληση των περικοπών του προϋπολογισμού. Τεράστιες περικοπές, 20% σε κάποιες χώρες. Στο Βέλγιο έχουμε πετύχει με τους στόχους μας, αλλά ένα τέταρτο του προσωπικού έφυγε, μειώθηκε σημαντικά ο προπολογισμό μας και βλέπουμε όμως ότι έχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα και πετυχαίνουμε τους στόχους μας και μπορούμε να συμμετέχουμε σε στρατιωτικές ε, επιχειρήσει στο εξωτερικό μετά από απόφαση σχετική της ε, κυβέρνησής μας και των κοινοβουλίων μας. Έχουμε πολύ σύγχρονο εξοπλισμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας ε, για το Δεκέμβριο, ότι με τις νέες επενδύσεις που γίνονται, καταρχάς θα πρέπει οι επενδύσεις αυτές να είναι σε νέα υλικά, να, είναι, έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και κατά προτίμηση να είναι διαλειτουργικές οι επενδύσεις. Γιατί βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου πραγματικά δεν χρειάζονται αλληλεπικαλύψεις. Πραγμάτων δηλαδή που υπάρχουν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σε στρατιωτικό πλαίσιο, πραγματικά θα πρέπει να δώσουμε τη δική μας έμφαση και θα πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ και αυτή είναι η ουσία αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και κάτι, ένα στοιχείο για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τη Συνόδου. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά την αναδιαμόρφωση του προπολογισμού. Έχουμε για το μέλλον πολλά σημαντικά επενδυτικά προγράμματα, πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ αναρωτιούνται ποιοι θα είναι οι διάδοχοι των F-16, των Eurofighter κτλ. και όλου του σχετικού εξοπλισμού. Τι θα κάνουμε. Βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν κάποιες ομάδες χωρών που συνεργάζονται. Ναι, πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει όχι μόνο για λόγους χρημάτων, αλλά για στρατηγικούς και λειτουργικούς λόγους. Άρα, τα κονδύλια και οι περικοπές δεν θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση, αλλά μπορούν να διαμορφώσουν και ένα νέο όραμα της πολιτικής άμυνας και σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης. Την ερώτηση έχω ε, επίσης να απαντήσω του Γερμανού συναδέλφου για το συνάδελφο 346. Για το άρθρο 346. Να σας πω αυτό που είπατε για τα θέματα επικυριαρχίας. Είναι πάρα πολύ σωστό. Νομίζω ότι το άρθρο 346 ωστόσο αποτελεί μια παγίδα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. για το κατά πόσο θα πρέπει να διαμορφώσει μια πιο αυστηρή στάση σε ό,τι αφορά το άρθρο 346. Νομίζω ότι αυτό αφορά μια βασική ρήτρα για πολλά κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαμορφώσει πιο αυστηρούς όρους Ιδάλλως θα δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υπάρχουν κράτη-μέλη στα οποία επιτρέπεται να μην το κάνουν, να μην υπακούν. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό έργο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα κοινά προγράμματα άμυνα και μετά να έρθω στο θέμα της EDA. Αυτή η υπηρεσία Ευρωπαϊκής Άμυνας. Δεν νομίζω πως είναι μια επιλογή ότι τίθεται το θέμα κατά πόσο πρέπει ε, να έχουμε περισσότερες επιλογές, περισσότερο προσωπικό για την υπηρεσία. Όχι. Ε, πρέπει να υπάρχει η πολιτική ε, πρωτοβουλία, ένα άνοιγμα, ώστε το, η υπηρεσία να μπορεί να έχει τις δυνατότητες να κάνει τη δουλειά της. Αν δεν κάνω λάθος, η υπηρεσία έκανε 140 προτάσεις μεταξύ των οποίων και αυτή που είναι η δυνατότητα ανεφοδιασμού, η δυνατότητα ανταλλαγή πληροφοριών κτλ. Αλλά ο σκοπός της είναι να κάνει πολλά περισσότερα. από όταν να είναι ένα σύνδεσμο για στρατιωτικές αγορέ. Έχει να πει για το όραμα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, αλλά πρέπει να έχει και το πολιτικό άνοιγμα να μπορεί να, να, να, αφήσουμε μάλλον τη δυνατότητα στην υπηρεσία αυτή να κάνει τη δουλειά της, που πιστεύω ότι κάνει υποδειγματική δουλειά και εξαιρετικό έργο. Εγώ στο ομιλία μου τόνισα αυτό το ρόλο και μετά από την εβδομάδα της Γάνδης είχαμε συμφωνήσει πως για το, την, τη μοιρασιά και την αμοιβαιότη πίση θα πρέπει η υπηρεσία να παίξει το ρόλο της. Γιατί πώς να το πω, είναι πάλι αυτή η παλιά ιστορία από το ποτηριού που το βλέπει κανείς μισογεμάτο ή μισοάδιο. Για μένα, με αυτή την, αυτή την υπηρεσία, το ποτήρι είναι μισογεμάτο. Υπάρχουν δυνατότητες πολλές Ίσως θα πρέπει να βάλουμε λίγη ζαχαρίτσα για να νοστιμήσει κάπως και το, το νερό που έχει μέσα το ποτήρι. Το Συμβούλιο που συνεδριάζει με σε επίσημο σχήμα. Έχει αλλάσει η μορφή, δηλαδή οι Υπουργοί Αμήνης τώρα συνεδριάζουν μόνοι τους κατά τις διάφορες προεδρίες. Πρόκειται για μια δομή που μεγαλώνει, αυξάνεται. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν έχει φτάσει ακόμα σε ενήλικο στάδιο. Έχουμε πάντοτε την εντύπωση πως δουλεύουμε όχι εν κενό ακριβώς, αλλά ότι η διασύνδεση με τα άλλα επίπεδα απόφασης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι εγγυημένη. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Οι υπουργοί αμήνης που συνεδριάζουν χωρίς οι συνάδελφοί τους των εξωτερικών υποθέσεων να είναι δίπλα τους, μπορεί να επιφέρει απώλεια παραγωγικότητας, για να μην πω απώλεια χρόνου. Ναι, βεβαίως να συνεδριάζουμε, αλλά αν είναι να συνεδριάζουμε για να μεταβάζουμε μετά ένα σημείο μας στους άλλους συναδέλφους, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι η θεσμοθέτηση θα ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Αλλά τότε αλλά με κάποιο τρόπο να υπάρχει, να μπορούμε να έχουμε επιρροή ε, στις ε, αποφάσεις που θα ληφθούν αργότερα. Αλλά είμαι υπέρ. Υπάρχει πιθανότητα το Συμβούλιο να μπορέσει να δώσει μια τέτοια ε, δυνατότητα. Ναι, κοιτάξτε, το συζητάμε τους μόνιμους εκπροσώπους. Ε, εγώ δεν είμαι υπέρ ε, τη ε, θαυματουργής μοιρασιάς ψωμιού στο Συμβούλιο. Όχι, έχουμε αρκετά επίπεδα λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν και παντού. Απλώ πρέπει να τα κάνουμε να λειτουργήσουν. Είναι θέμα στάσης και βούλησης. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί με εντυπωσίασε αυτό που είπατε για το ότι ναι, αν θέλουμε να έχουμε πραγματική ποιοτική πρόοδο, θα πρέπει μεγάλες χώρες μεταξύ εισαγωγικών, δηλαδή Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία, να παίξουν το παιχνίδι, να, να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Εσείς που προέρχεστε από ένα light-minded, μικρότερο δηλαδή κράτος μέλος, ε, αυτό που με εντυπωσιάζει πολύ είναι ότι το Βέλγιο είναι πολύ παρόν σε όλες τις επιχειρήσεις. Είτε είναι ο συνασπισμός των προθήμων, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Βέλγιο συμμετείχε και στις επιχειρήσεις στη Λιβύη και στο Μαλί. Μας μπορείτε να μας πείτε για τις ε, μικρές αλλά σημαντικές δυνατότητες και επί των οποίων μπορούμε να στηριζόμαστε στο Βέλγιο. Έχουμε εξειδικευτεί όπως ε, θέλουμε να γίνουμε σαν τις τρεις μεγάλες χώρες είναι κάτι που θέλουμε μετά από την πολιτική συνένεση να το κάνουμε αμέσως, αμέσω. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα όπως κάναμε στο Αφγανιστάν που πήγαμε. Και στην Αταλάντη επίσης και στις άλλες επιχειρήσεις που έγιναν στις ακτές της Δυτικής Αφρικής και εκεί ήμασταν παρόντες. Στη Λιβύη, Unified Protect, εκεί ήταν το πιο κλασικό παράδειγμα και για ιστορικούς λόγους επίσης ε, στην Προνιγκοσλαβία λίγες στον Λίβανο και επίσης στην ε, Αφρική. στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στο Κονγκό. Εκεί που είχαμε τις επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Ανατολικά στη χώρα εκείνη, στο εντολικό τμήμα, πολύ σημαντικό το τι έγινε εκεί και αυτό δείξει ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε σε διαφορετικά εδάφη, σε διαφορετικού χαρακτήρα αποστολές, πάντοτε υπό την υγίδα κατά προτίμηση του ΟΗΕ. Σχετικά τώρα με τη Συρία, Είχε γίνει συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Και βέβαια το, το, το συζητούσαμε, ήταν αλλιώ η διεθνή συγκυρία πριν από δύο-τρει ε, εβδομάδες, αλλά δεν θα καλά γίνει μια σύνοδος υπουργών εξωτερικών στη Νέα Υόρκη. Κανονίστηκαν οι προϋποθέσεις. Οπότε και αποφασίστηκε και για το Βέλγιο ε, λόγω συγκεκριμένων δυνατήτων και γνώσεων σε σχέση με τα χημικά όπλα. Οπότε αποφασίστηκε η ενδυνάμιση συμμετοχή μας σε ενέργειες κατά των χημικών όπλων στη Συρία. Για ιστορικούς λόγους υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις πάντοτε, αλλά δεν μπορούμε να μιλούμε για αλληλεγγύη και για διαλειτουργικότητα. Δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα στους άλλους ε, όταν μας ζητείτε κάτι και εμείς αρνούμεθα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και στο το και σε άλλες επιχειρήσεις υπό αλληλεγγύδα ας πούμε σε επιχειρήσει που έχει τον διευθύνοντα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέμε ότι να έρθουν ε, ε, να έρθουν όποιοι θέλουν και κάποιοι πάντοτε να διστάζουν. Δεν είναι σωστό. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να ανήκει σε έναν φορέα και όταν ε, καλείται να βοηθήσει να μην συμμετέχει. Δεν μπορεί να βγάζουν το φίδι από την τρύπα πάντοτε οι ίδιοι. Αλλά και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ξέρετε, και εκεί θα πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας. Ζήτησαν, είπα, να συμμετάσχουμε στην κατανομή του βάρους, στην χρηματοδότηση, ως, σε ό,τι μας αναλογεί για την ασφάλεια. Αυτό είναι 100% κατανοητό. Άρα, ετοιμαστείτε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να συζητηθεί αυτό στην ε, Υποπιτροπή Άμυνας. Αυτά ήταν τα κατηγορητικά σας σχόλια, κύριε ε, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας. Βέβαια εννοείται ότι σας περιμένουμε να ξανέρθετε όποτε μπορέσετε και κυρίως ε, μετά τη διάσκεψη κορυφής. Ελπίζουμε να μην κατησχίσουν μόνο τα οικονομικά, τα πολιτικά εκεί. Να σας περιμένω τέλο πάντων ε, του χρόνου στο πρώτο τρίμηνο για να δούμε πώς έχει κατάσταση. Πολύ πολύ πολύ μικρό διάλειμμα για να συνοδεύσουμε στην έξοδο τον Υπουργό και στη συνέχεια θα συζητήσουμε για την κατάσταση στη Συρία. Ευχαριστώ.

σε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 Θα μιλήσουμε για την κατάσταση στη Συρία που όπως γνωρίζετε είναι εξαιρετικά μεταβλητή ε, ε, από στρατιωτικής και διπλωματικής άποψης. Εμείς βέβαια δεν ε, σκοπεύουμε να εξαντλήσουμε τώρα εδώ το θέμα σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στη Συρία και στο φάκελο Συρία γιατί στη Νέα Υόρκη οι εξελίξεις συνεχίζονται. Αυτό που θα ήθελα να κάνουμε είναι να μιλήσουμε για την κατάσταση στη Συρία και ίσως τι σημαίνει αυτό σε θέματα αμήνης στρατιωτικά, δεδομένου το ότι έγινε στις 21 Αυγούστου. Η υπόθεση μιας στρατιωτικής επέμβασης ε, έχει για την ώρα ανασταλεί, αλλά δεν έχει ακυρωθεί δεν είναι κάτι που να έχει τελείω δηλαδή ξεπεραστεί. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι μπορεί και να ξαναχρειαστεί να μιλήσουμε για στρατιωτική επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό μένει στο πλαίσιο του δυνατού, του πιθανού. Και υπάρχουν κάποιες ε, ε, εντυπώσεις όσον αφορά <coughs> τα όσα συμβαίνουν επί τόπου. Καλέσαμε δύο εμπειρογνώμονες και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Δεν είναι και εύκολο γιατί για τη Συρία <laughs> πιο πολύ προβλέψεις κάνουμε ε, και υποψίες έχουμε παρά συγκεκριμένα γεγονότα και γνώσεις για το τι ακριβώς τρέχει επί τόπου. Στα αριστερά μου, ε, Julian Barnes Dassey, που είναι πυρογνώμονες ε, και εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων ε, και η έκθεση που έγραψε για τη Συρία μου φάνηκε πολύ σκόπιμη και πιο αριστερά ο κύριος Ζαν Πασκάλ Ζάντες που είναι ερευνητής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Μελετών για την Ασφάλεια, δράζει το Παρίσι, είναι ειδικό για τις εξοπλισμούς και ιδιαίτερα για τα χημικά, βιολογικά και πυρηνικά όπλα. Ιδιαίτερα χρήσιμος λοιπόν για να μας πείτε και τα όσα συμβαίνουν στη Σύρια αυτή τη στιγμή. Μάλιστα θα σας δώσω πρώτα το λόγο κύριε Ζαν Πασκάλ Ζάντερς και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπάνς Ντάση. Κύριε Πρόεδρε, Εξαιρετικά μέλη της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και ε, Άμυνας και Ασφάλειας ε, έχω την τιμή να σας μιλήσω για τα χημικά όπλα και την αφοπλισμό στη Συρία. Από ό,τι κατάλαβα διάφορες πρόσφατες εισηγήσει μου σας έχουν δοθεί ως βάση για τα όσα θα πω και εγώ θα περιοριστώ στο να τονίσω κάποια βασικά θέματα. Στις 21 Αυγούστου ο κόσμος ξεκίνησε να λειτουργεί με τα νέα μεγάλων ε, ε, ε, χτυπημάτων στην περιοχή Γκάουτα της Δαμασκού. Εκατοντάδες κόσμος έχασε τη ζωή του από τις ε, επιπτώσεις δηλητηριωδών αερίων και πολλοί άλλοι θα υποφέρουν από τις μακροπρόθεσμες ε, επιπτώσεις του αερίου που χρησιμοποιήθηκε που τώρα ξέρουμε ότι ήταν το Σαρίν. Από τα τέλη του 2012 υπήρξαν διάφοροι ισχυρισμοί για τη χρήση χημικών όπλων αλλά καμιά από αυτούς δεν είχε επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Αν και αναφέρθηκαν θάνατοι και άλλα ατυχή και άλλα θύματα, η συνολική εικόνα ποτέ δεν οδήγησε στο να πιστέψουμε ότι γινόταν χημικό πόλεμο. Ωστόσο, η φύση τη επίθεση στην περιοχή Γκάουτα έφερε με σημαντικό τρόπο από του υπόλοιπου ισχυρισμού. Η τα παράλληλα χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, ο αριθμός των θυμάτων και η πυκνότητα των τοπικών αναφορών, δηλαδή ε, οι μαγνητοσκοπήσεις, εικόνες αλλά και οι αναφορές των ε, επιτόπου μαρτύρων, Όλα αυτά ε, τη σοβαρότητα του θέματος. Αυτή τη στιγμή είμαι σχετικά ικανοποιημένος γιατί οι επιθέσεις στην περιοχή Γκάουτα δεν μπορούσαν να είχαν γίνει από τους ε, Η Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ παρουσίασε στις 16 Σεπτεμβρίου. Το έγγραφο ανεξάρτητα επιβεβαιώνει τη χρήση χημικών στον ε, φίλιο της Συρίας. Ε, είναι αδιαφεσβήτητο το συμπέρασμα ότι όλα αυτά βασίζονται σε πάρα πολλά δείγματα, στις συνδεύξεις με τα θύματα, στην έρευνα των υπολοιμάτων των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν και σε αναλύσεις εργαστηριακές. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτές τις επιθέσεις που δεν αποσαφηνίζει απόλυτα η έκθεση του ΟΗΕ. Ανάμεσα στα θέματα που πρέπει ακόμα να αναλυθούν, πέραν πάσης υποψίας, αποτελεί το είδος των συστημάτων ε, εκτόξευσης και, σε ποιον ανήκουν όλα αυτά, ανάλυση επίσης και ποιότητα, της ποιότητας του σαρίν και κατά πόσο αυτό το αέριο έχει φτιαχτεί βιομηχανικά ή ε, βιοτεχνικά και ούτω καθεξής. Τώρα, οι εκτιμήσεις των, ε, της ε, αντικατασκοπίας ε, για τις επιθέσεις στην ΚΑΟΤΑ από πλευράς Γαλλίας και Ηνωμένων Βασιλείου αλλά και ΙΠΑ βασίζονται εν μέρη σε προηγούμενους ισχυρισμούς για τη χρήση χημικών ώστε να θεσπιστεί ένα σχήμα συμπεριφορά για την Συριακή κυβέρνηση. Ωστόσο, οι μαρτυρίες, οι ενδείξεις αυτές είναι λιγοστές και πολλές χώρες αυτές δεν έχουν δώσει όλες τις λεπτομέρειες ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα να μπορέσει να τις αναλύσει. Τους τελευταίους μήνες έχω επανειλημμένως προειδοποιήσει ότι το να πουλάμε πολύ τις περιορισμένες αποδείξεις που έχουμε στη διαθεσή μας είναι επικίνδυνο γιατί τα στοιχεία εξυπηρετούν βασικούς στόχους σε αυτή την περίπτωση η στρατιωτική επέμβαση. Ε, οι γελιοποιούνται ως και οι πολιτικοί καταγράφουν τα στοιχεία τα οποία έχουν περισσότερη αξία ε, ως αποδείξεις από ό,τι ε, πραγματικά έχουν. Όλα αυτά λοιπόν χρησιμοποιούνται ως λογική αμφιβολία και αυτό επιτρέπει και στη Ρωσία να ε, συνεχίζει να στηρίζει την Συριακή κυβέρνηση. Η Ρωσία και η ΙΠΑ επέτυχαν μια συμφωνία για την ε, καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας στη Γενέβη της 14 Σεπτεμβρίου. Η Συρία ανακοίνωσε ότι θα γίνει το 190ο κράτος που θα υπογράψει τη Σύμβαση Περιχημικών στις 14 Οκτωβρίου. Είναι η πρώτη περίπτωση ε, που θα χρησιμοποιηθούν όλα τα σχετικά, οι σχετικές προβλέψεις ε, της ε, σύμβασης. Δηλαδή το εκτελεστικό συμβούλιο θα πρέπει τώρα να θέσει προθεσμία ε, απότατη συμφωνία για την καταστροφή των χημικών όπλων. Από όσο γνωρίζω αυτή η απόφαση ακόμα δεν έχει ληφθεί, εκκρεμεί και τη απουσία της είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε κατά πόσο είναι εφικτές αυτές οι προθεσμίες που περιλαμβάνονται στις συμφωνία πλαίσιο. Η σχέση ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ενός κράτους που έχει συνυπογράψει τη συμφωνία και τα συγκεκριμένα αιτήματα στο πολιτικό έγγραφο ε, είπα Ρωσία θα πρέπει να μεταφραστούν σε νομικώς δεσμευτική και άρα ε, ε, δυνατόν να επιβληθεί η συμφωνία. Είναι σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα για κεντρικό ρόλο για δύο ε, διεθνείς ε, οργανισμούς, τον Οργανισμό για την ε, Απαγόρευση των Χημικών Όπλων και, τους, και τον ΟΗΕ. ο αφοπλισμός θέλει να, να αφαιρέσει μια διακριτική κατηγορία όπλων από το στρατιωτικό δόγμα μιας πολιτικής οντότητας. Η καταστροφή των όπλων είναι μία πτυχή, ενώ το να πάψει κανείς να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ή να αναπτύσσει τέτοιου είδους όπλα είναι το πιο σημαντικό δεν γίνεται πλέον δοκιμή στα πυρομαχικά, δεν υπάρχει κατάρτιση, εκπαίδευση των ε, στατευμάτων για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Για, ε, εν τω μεταξύ, οι επιστήμονες, οι μηχανικοί και οι τεχνικοί χάνουν τη τεχνογνωσία τους ώστε να βελτιώνουν διαρκώς ε, το σχεδιασμό όπλων και τις δυνατότητες παραγωγής. Εάν ε, το δόγμα, από μια, ε, μάλλον ε, ένα συγκεκριμένο όπλο από το στρατιωτικό δόγμα σημαίνει ότι μειώνονται οι πιέσεις όσον αφορά την εξέλιξή του και την χρήση του. Επίσης, ο αφοπλισμός σημαίνει πρόληψη των πολέμων. Συμβάλλει στην ειρήνη και την ασφάλεια αυτό συνέβη με τα χημικά όπλα κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 30. Ακόμα και αν ξεσπάσει πόλεμο, ο αφοπλισμός εμποδίζει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μάχη ή σε μια κλιμάκωση των εχθροτήτων. Εάν μεταφραστεί στη Συμφωνία Πλαίσιο ΙΠΑ Ρωσία, το να αναγκαστεί η Συρία να εγκαταλείψει το χημικό τη οπλοστάσιο θα, θα, θα σημάνει ότι δεν μπορεί πια να ε, υπάρξει περίπτωση γκάουτα στο μέλλον. Εάν η Συρία όντω συνυπογράψει τη συμμετοχή τη ε, στη σύμβαση, η Ρωσία και η ΗΠΑ θα έχουν καταστήσει την, το χημικό αφοπλισμό της Συρίας μια παγκόσμια μακρόχρονη ευθύνη και όχι μια ad hoc λύση σε ένα πιεστικό πρόβλημα. Εάν επιτύχει, η ευρύτερη συμβολή της Συμφωνίας Πλαισίου στον αφοπλισμό μπορεί να είναι η εισαγωγή μιας νέας δυναμικής στην αποκαλούμενη διαδικασία του Ελσίνκη, ώστε να συγκληθεί μια συνεδρίαση για την ε, καταστροφή των μη συμβατικών όπλων στην Μέση Ανατολή, όπως ζητήθηκε από το τελικό έγγραφο της ε, της ε, διάσκεψης για την αναθεώρηση της συνθήκης περί μη εξάπλωσης των μη συμβατικών όπλων. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις στρατηγικές σχέσεις ανάμεσα στην Αίγυπτο, την, το Ισραήλ και την Συρία, θα πρέπει να ξαναδούμε τι ισχύει τόσο όσον αφορά τις δογματικές σχέσεις ανάμεσα στα απλοστάσια τους, αλλά και τη συμμετοχή τους στις, στη σύμβαση, στις συμβάσεις και βιολογικών όπλων. Τώρα, ε, το, το, θέμα του Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα ίσως χρειάζεται διαφορετική δυναμική. Τα όσα μας στάνουν από τις συναντήσεις του ΝΟΙΕ είναι θαρρυντικά και οι Ιρανικές ε, πρόσφατες εκλογές μπορεί να αποτέλεσαν ε, το σημείο καμπής ώστε να σπάσει το αραστεγές κάλυμα του Ιράν και απομόνωσή του από τον υπόλοιπο κόσμο. Και όπως πρόσφατες αναφορές στον τύπο λένε, μπορεί επίσης να συμβάλλει ε, το Ιράν για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Μπορούμε να φανταστούμε όμως αυτή τη δυναμική ε, με λίγες ε, τιμωρητικές επιθέσεις αεροπορικές να γίνονται πριν από λίγες εβδομάδες. Μόνο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και τώρα η εισήγηση λίγο διαφορετική από τον κύριο Μπάνς Ντάση. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου κάνετε την τιμή να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για τη Συρία σήμερα. Θα είμαι αρκετά σύντομος για να μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση μετά. Να σας δώσω λοιπόν κάποια αρχικά ε, θέματα σε ό,τι αφορά την ευρύτερη κατάσταση στην Συρία και την πολιτική δυναμική για την ε, διπλωματική και παρεμβατική ενδεχόμενη πορεία. Να ξεκινήσουμε αναφέροντας πώς έχει κατάσταση επί τόπου. Είναι σαφές ότι παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι μάχες, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καμία πλευρά δεν μπορεί να κερδίσει. και δεν φαίνεται να αλλάξει αυτό σύντομα. Το καθεστώς εξακολουθεί να έχει έλεγχο σε κάποιες ε, πόλεις ε, στην πρωτεύουσα, στις μεγάλες πόλεις της Συρίας, αλλά και οι αντάρτες ε, έχουν τον έλεγχο από το βόρειο μέχρι το ανατολικό κομμάτι της χώρας και αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση σε όλη την Συρία σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Άρα, το καθεστώς το εφιστάμενο είναι και η κυβέρνηση είναι ενιαίο, δυνατό, παρά το γεγονός ότι οι αντάρτες ε, αποκτούν όλο και πιο πολύ δύναμη και δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιος ε, κατακριματισμός που θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα ε, εγκαταλείψουν τις θέσεις τους. Και επίσης ε, το γεγονός ότι έφυγε ο Αλχαμπίμπα από την άμυνα μάλλον θα ενισχύσει την θέση της κυβέρνησης. Δεν υποδεικνύει ότι υπάρχει εσωτερικός κατακαιρματισμός από πλευρά των ανταρτών. Θεωρώ ότι η κατάσταση δυσκολεύει και πάει αντιμετωπίζουν όλο και πιο πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την ενιαία τους χαρακτήρα ως πολιτική δύναμη παρά το γεγονός ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση από πλευρά στρατιωτικής τελευταίες εβδομάδε βλέπουμε ότι υπάρχει διχόνοια. Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά για το μέλλον. Βλέπουμε ε, αυξημένες ε, διαμάχες μεταξύ των πιο ακραίων στοιχείων και αυτό το βλέπουμε και στον τύπο κάποιες απόπειρες ε, να επισέλθουν Κούρδοι στα βασικές πολιτικές ομάδες στο εξωτερικό και αυτό υποδεικνύει το ότι το PRD αποξενώνεται και πάει και επίσης αύξηση του εξτρεμισμού το 50% των άνταρτων σήμερα προσυπογράφουν σε κάποιο ακραίο ισλαμιστικό ή σε ακραία ισλαμιστική ιδεολογία σύμφωνη με μια μελέτη και χτες δημοσιεύθηκε μια δήλωση όπου ουσιαστικά προσυπογράφουν αυτές, ε, αυτό το, το γεγονός ότι α, ανήκουν στις Ισλαμιστικές ομάδες και ότι δεν ε, υποστηρίζουν το SNC. Το σενάριο το οποίο χρησιμοποιούν οι Ρώσοι είναι ότι υποστηρίζονται όσο πιο πολύ οι τσιχαντιστές και όσο προχωράει ο καιρός όλο και πιο πολύ αναδεικνύεται αυτό το σενάριο Ασάντ θεωρείται ότι είναι το αίτιο του σενάριου αυτού, αλλά παραδόξως αποτελεί και την οικολογία κατά του σενάριου αυτού. Τώρα, έγινε κάποια συζήτηση για θέματα παρέμβασης. Να έχουμε υπόψη μας ότι ό,τι έγινε τονίζουν ότι υπάρχει έλλειψη προθυμίας από πλευράς της Δύσης για να παρέμβουν πραγματικά, αλλά και βασικά την έλλειψη των ε, σωστών και απαραίτητων δυνάμεων. Μία παρέμβαση θα έχει συμβολική σημασία, αλλά ακόμα και αν είχε κάποια αντίκτυπο σε ό,τι αφορά ε, τη χρήση χημικών όπλων, θα είχε στρατηγική σημασία ε, επιτόπου σε ό,τι αφορά τη μάχη. Τα χημικά όπλα είναι ασφαλώς πάρα πολύ σημαντικά και συμβολική σημασία, αλλά παρόλα αυτά εκπροσωπούν ένα 1% μόνο των συνολικών θανάτων και σε ό,τι αφορά την απειλή για την Ευρώπη, ναι, τα χημικά όπλα αποτελούν μια απειλή, αλλά ο τζιχαντισμός και η τζιχάτα αποτελεί νομίζω ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη απειλή. Ούτε θεωρώ ότι ένα τέτοιο αντικίνητρο, ένα φόβητρο θα μπορούσε να λύσει την πολιτική κατάσταση. Χρειαζόμαστε σε καμία περίπτωση δεν ε, μπορούμε να πούμε ότι στην παρούσα φάση μία από τις δύο πλευρές είναι δεθμένη να κάνει πολιτικές κινήσεις ε, βασμού. Οι ε, επαναστάτες από πλευράς τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύουν να συνεχίσουν διαπραγματεύσεις με το καθεστώς. Και αυτό νομίζω σε τελική ανάλυση θα χρειαστεί πολιτική συμβιβασμό προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαμάχη και ο Ασάντ και η υποστήριξη της Εσμπολά του Ιράν θεωρούν ότι αυτό αποτελεί ε, ένα σπρώξιμο προς το Ιράκ και ότι η Συρία βασικά έχει να κάνει με την αλλαγή του καθεστώτος στην Τιχεράνη και είναι σαφές ότι η δυτική παρέμβαση θα ήταν πάρα πολύ περιορισμένη σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των δυναμικών αυτών και κατά πάσα πιθανότητα θα πυροδοτούσε τους φόβους ε, των μειονοτήτων στη Συρία που φοβούνται όλο και πιο πολύ ότι η κίνηση, το κίνημα των Σουνιτών, ε, των Ισλαμιστών στην Συρία θα τους απειλήσει και δεν θα έχουν μέλλον αν ε, η Δύση τους υποστηρίξει. Η πραγματικότητα είναι ότι ο μοναδικός τρόπος ε, που θα μπορούσε να έχει αντικτύπω μια στρατιωτική παρέμβαση είναι εάν πρόκειτο για μια μεγάλη έκτασης παρέμβασης που θα έφερε τέλος στην ε, διαμάχη. Η μοναδική λύση λοιπόν θα ήταν μια παρέμβαση τύπου Ιράκ, το οποίο προφανώς δεν το εξετάζουμε σε ό,τι αφορά και τον κίνδυνο που θα ενείχε. Και πόσο μάλλον τι θα γινόταν μετά. Για το κατά πόσο θα υπήρχε δομή για μια Συρία μετά τον Ασάντ. Το πιο πιθανό σενάριο θα ήταν ένας νέος εμφύλιος πόλεμος, μιας και φαίνεται ότι κατακαιρματίζεται και το μέτωπο των ανταρτών μεταξύ των πιο ακραίων και των πιο μετριοπαθών στοιχείων. Η απειλή νομίζω ότι έχει να κάνει με το άνοιγμα ενός τέτοιου διπλωματικού παράθυρου. Αυτό είναι θετικό. Η απειλή άσκησης ε, βίας, η απειλή παρέμβασης. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία και η στάση της έχει να κάνει με μια τέτοια μετάθεση και αλλαγή των δυνάμεων επιτόπου. Μόλις ήρθα από μια επίσκεψη στη Ρωσία. Η Ρωσία φοβάται ότι αυτό θα θέσει ένα προηγούμενο το οποίο θα ξεκινήσει στη Λιβύη σε ό,τι αφορά το, τη μονομερής παρέμβαση της Δύσης άσχετα με το τι θα γίνει με τους αντάρτες και την νίκη τους σε ό,τι αφορά τα χημικά όπλα τώρα. Μία τέτοια δράση μπορεί να έχει αποτελέσματα μόνο αν υπάρχει ευρεία πολιτική στήριξη. Θα χρειαστούν και χειρίες επιτόπου. Θα πρέπει να καταστραφούν όλα τα όπλα αυτά. Αυτό θα χρειαστεί μια ανακοχή Άρα θεωρώ ότι υπάρχει μια ευκαιρία να προχωρήσουμε και να ακολουθήσουμε ένα δρόμο, το μοναδικό δρόμο ειρήνευσης και συμφιλίωσης, προκειμένου και οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Δεν μπορούν οι εντάρτες να νικήσουν απόλυτα. Θα χρειαστεί να κλείσουν συμφωνίες, θα πρέπει το Ιράν να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να διαπραγματευτούν το θέμα και της μοίρα του Ασάντ και αυτό θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα, αν θέλετε, των συζητήσεων, όχι ένας όρος που θα δεθεί εκ των προτέρων. Και... Ο Ασάντ, ε, είτε το θέλουμε είτε όχι, ε, έχει κερδίσει ένα, μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και οι αντάρτε θα πρέπει να το δεχτούν αυτόν. Άρα δύο πράγματα θα πρέπει να γίνουν τώρα. Καταρχάς, ότι ο συμβιβασμός αυτός ε, πέρα από το τι πιστεύουν οι Ρώσοι και οι Ιρανοί θα πρέπει να γίνει και ότι υπάρχει πίεση και σε, στις δύο πλευρές ότι μιας και δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ίδια κατεύθυνση και την ίδια πορεία θα αναγκαστούν να διαπραγματευτούν. Και θα πρέπει η Ευρώπη να πιέσει προς την κατεύθυνση αυτή ότι δεν υπάρχει απόλυτη νίκη. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τα ανθρωπιστικά ζητήματα σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, σε ό,τι αφορά τις ροές προς το Λίβανο. Η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί πολύ περαιτέρω. Δεν υπάρχει, θεωρώ, ελπίδα για να νικήσει κάποιος ξεκάθαρα και οι δύο πλευρές πλέον εξαρτώνται από εξωτερική υποστήριξη από τους Ρώσους, από τους Ουρανούς, από τη Χεσμολά, από την Τουρκία, τις χώρες του κόλπου, από πλευράς των ανταρτών, πολιτικός, ε, οικονομικός αλλά και στρατιωτικά. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια τεθνή έκκληση για την έβρεση συμβιβασμού προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση στη Συρία προκειμένου να καταλάβουν και οι δύο πλευρές ότι δεν υπάρχει προοπτική νίκης. Προς το παρόν, οποιαδήποτε συζήτηση για παρέμβαση της δύση ε, πυροδοτεί αυτή την ελπίδα απόλυτης νίκης, χωρίς να αλλάζει όμως με κανένα τρόπο τη δυναμική της κατάστασης. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξουμε μια διεθνή πολυμερή διαδικασία έβρεση συμβιβασμού συμφωνίας παρά να ακολουθήσουμε ε, μια απόλυτη διαδικασία διαπραγματεύσεων ή μια απόλυτη νίκη που θα προαπαιτεί ότι δεν θα συμμετέχει ο Ασάντ, ότι δεν θα εμπλεχθούν ξένες δυνάμεις και το καθεξής. Ο Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισήγησή σας, η οποία νομίζω ότι θα προκαλέσει πολλές ερωτήσεις και αντιδράσεις. Εγώ από πλευράς μου έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη έχει σχέση με την καταστροφή των χημικών. Αυτή θα πρέπει να γίνει συνενετικά, έτσι φαίνεται, και να δούμε με ποιο τρόπο ακριβώς και από την άλλη μεριά θα, θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, όπως το παρελθόν έχει γίνει. Πώς ακριβώς όμως θα καταστραφούν τα όπλα αυτά, γιατί πολλά κυκλοφορούν λένε ότι θα πρέπει να συγκροτήσουμε κάποιες εξειδικευμένες βιομηχανικές μονάδες επιτόπου τόσο ώστε να προβούν στην ασφαλή καταστροφή ή ότι θα πρέπει να καταστρέψουν αυτά τα χημικά εκτός Συρίας. Συγκεκριμένα πώς θα προχωρήσουμε τώρα όσον αφορά ε, τα, τα, τα πλήγματα, τα τιμωρητικά ε, είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι μπορούμε να χτυπήσουμε τις εγκαταστάσεις των ε, χημικών τις εγκαταστάσεις τέλο πάντων εκτόξευση των χημικών πυράβλους. Πώς θα γίνει αυτό, ή δεν μπορεί να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Επίση, ε, Στις Βεξέλλες επίσης ε, υπάρχει συζήτηση όσον αφορά την άρση του εμπάργου ε, για την πώληση όπλων στους αντάρτες οπότε τι γίνεται με τον οπλισμό του, γιατί αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ε, δείτε την εντύπωση ότι υπήρχαν κάποιοι εκεί οι οποίοι πολεμούσαν με πρωτόγωνα όπλα κατά ε, ενός στρατού πάρα πολύ σύγχρονο. Εκτός βέβαια από τους ε, πυράβλους εδάφους αέρας, ότι η αντιπολίτευση είχε ε, κάποια όπλα από τις χώρες του κόλπου. Τι είναι αυτό, κάτι σαν ένα μυστήριο πώς βρέθηκαν με αυτά εσείς τι λέτε, τι οπλισμό έχουν οι ε, στασιαστές, οι επαναστάτες, η αντιπολίτευση και ποιος τους δίνει τα όπλα. Πάντως να μην μακρηγορήσουμε διότι έχουμε ένα 40 και θα ήθελα επομένω να δώσουμε τον χρόνο στους ε, εισηγητές να μας παντήσουν για την καλύτερα. Κύριε Καταρχάς, με τη σειρά μου να καλωσορίσω και να συγχαρώ τους ομιλητές μας οι οποίοι πραγματικά κατάθεσαν δύο πολύ ολοκληρωμένες θα έλεγα προτάσεις. Η δική μου θέση είναι παρέμβαση πολιτική για τα γεγονότα γύρω από την Συρία και θεωρώ πολύ σημαντικό και το χαιρετίζω την επίτευξη συμφωνίας για την ουδετεροποίηση καταστροφή των προστασίου χημικών όπλων στη Συρία. Χαιρετίζω επίση ότι η Συρία προσχωρεί στην Διεθνή Συμφωνία για τα Χημικά Όπλα, κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η συμφωνία θα μειώσει, πρέπει να μειώσει σίγουρα τον αριθμό των θυμάτων του εφηλίου και βέβαια γιατί ταυτόχρονα αποφεύγεται μια στρατοτική επίθεση κατά της Συρίας που θα είχαμε θύματα, βία, τρομοκρατία, πιθανότατα πέρα από τα σύνορα της Συρίας, στον αραβικό κόσμο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αστάθεια τρομοκρατία αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κράτη-μέλη όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Βουλγαρία είναι δυστυχώς περισσότερες τροτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι μια αλήθεια. Αυτές οι χώρες έχουν ήδη σοβαρά προβλήματα υποδοχής μεγάλου αριθμών Σύριων προσφύγων. Παραδείγματο χάρη η Βουλγαρία υπέβαλε διαμαρτυρία στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών στι 24 του Σεπτέμβρη, διότι αδυνατεί να υποδεχθεί πρόσφυγε Το ίδιο ισχύει για την Κύπρο και την αλήθεια. Και την Ελλάδα, μια επίση αλήθεια. Είναι αναγκαίο λοιπόν να εξευρεθεί λύση, τονίζω, με διπλωματικά, με πολιτικά μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερο συμφέρον ως κύριος γείτονας της, της Μέσης Ανατολής και πρέπει να συνεχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες για την ειρήνη που θα αποκατασταθεί σταθερότητα στην περιοχή, να διαθέσει και άλλα μέσα και άλλη οικονομική βοήθεια για τους πρόσφυγες να περιορίσει, να περιορίσει την ανθρωπιστική καταστροφή. Και η πρόταση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> επιτέλους <clears throat> θα πρέπει να αυτονομηθεί και όχι να ακολουθεί τις Ηνωμένε Πολιτείες. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται, το τονίσαμε πάρα πολλές φορές, σαν μικρός αδερφός. Να πάρει πρωτοβουλίες ανεξάρτητα από τους στόχους, της επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών που πολλές φορές είναι διαφορετικοί οι στόχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να επιμείνει καθαρά στην εφαρμογή της σύμβασης του εμπορίου όπλων έτσι θα περιοριστεί ο συνεχής εξοπλισμός των τσιχαδιστών μέσων Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας. Να υπάρξει πίεση προς αυτές τις χώρες να σταματήσουν οι εξοπλισμοί αυτοί και βέβαια το όλο θέμα θα πρέπει να λυθεί με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ειρήνη θα φέρει σταθερότητα. Ο πόλεμος δυστυχώς την καταστροφή. Ευχαριστώ. Merci, Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ενημέρωση και επίσης για το κείμενο το οποίο διανύμεται και είναι ενδεχομένω πιο χρήσιμο. Σας ερωτώ, πώς αποτιμάτε το ρόλο της Ρωσίας, διότι ξέρουμε ότι εξοπλίζει το καθεστώς Άσαντ η Ρωσία. Επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία έδωσε χημικά όπλα ή τέλος πάντων τα συστατικά για την κατασκευή τους. Δεν έχει καταστρέψει τα δικά της ε, χημικά η Ρωσία. Δόθηκε παράταση για αυτή την ενέργεια. Πάντως νιώσαμε ανακούφιση όταν ε, απετράπη η παρέμβαση της νέας κοινότητας και ότι δεν θα υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση επιτόπου. Αλλά για πέστε μας για τα χημικά. Πώς θα μπορούσαμε να τα ανακαλύψουμε, πώς θα μπορούσαμε να τα καταστρέψουμε εκεί. Υπάρχει αρκετό εξειδικευμένο προσωπικό. Γιατί μου είπαν ότι η περίπου 120 ειδικού, που όμως βρίσκονται εγκατασπαρμένοι σε όλο τον κόσμο. Τώρα για την απομακρυνσή τους. Είναι σχεδόν αδύνατο κανείς να ανακαλύψει που βρίσκονται χωρίς να πέσουν στα χέρια των ε, ακραίων ενόπλων. Συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί είναι το εξής. Ε, έχουμε την κόκκινη γραμμή του Ομπάμα, από την οποία επανεχώρησε. Όμως ε, έχουμε την κόκκινη γραμμή του Πούτιν που υπεραμείνεται του Άσαντ. Και έτσι ο Άσαντ εξασφάλισε τη θέση του των διαπραγματεύσεων και κέρδισε χρόνο. Άρα, ερωτώ, τι τεχνικές δυνατότητες υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε τα χημικά και να τα καταστρέψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Κύριε Κρόμπεργκ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσε οι εισηγήσει. Συμφωνώ με την δυναμική που έχει αναπτυχθεί, όπως την εξηγήσατε. Είναι ενδιαφέρον το ότι τώρα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα χημικά και θα μπορούσε να υπάρχει με αφορμή την αντιμετώπιση αυτή μια διάσκεψη για την Μέση Ανατολή γενικότερα. Να έχουμε επομένω την αντιμετώπιση και την διάσκεψη αυτή από τη βάση τη Σύμβαση για τα Οπλομαζική Καταστροφή. Βέβαια, είπα και η Ρωσία τα συμφώνησαν. Η Συρία προσυπέγραψε τη σχετική σύμβαση για τα χημικά. Ακόμα όμως, ακόμα υπάρχουν προβλήματα. Παγίδες, εν δυνάμει. Ένα χρονοδιάγραμμα. Τζούλιαν, θα μπορούσατε να μας πείτε ποιοι είναι οι κίνδυνοι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη διαδρομή. Πού ελοχεύουν αυτοί οι κίνδυνοι. Πώς να ετοιμαστούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Λέζινγκ. Ναι, θα ήθελα και εγώ καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή παρουσίαση και συνοπτική. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση του σενάριου, του τι θα σήμαινε δηλαδή μια παρέμβαση, τι αντίκτυπο θα είχε. Και το παράδειγμα του Ιράκ αναφέρατε, καλό και αυτό. Τώρα λοιπόν μπορούμε να δούμε πού οδήγησε η δράση μας, τώρα μόλις Βλέπουμε ότι τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν, αλλά ότι το αποτέλεσμα ήταν χιλιάδες νεκροί επιπλέον και μια αποσταθεροποίηση της χώρας ολόκληρης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ καλό σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα και τα πορίσματα, ότι κοιτάμε ποιος θα κάνει τι και πότε. Δεν έχει αποδειχτεί αδιαφυσβήτητα από τις ε, εμπρεγνώμονες ε, τα θέματα αυτά. Και είναι σημαντικό το τι θα έπρεπε να γίνει. Τι θα έπρεπε να γίνει. Ακόμα και αν το καθεστώς ε, Ασάντ είχε αναστείλει τη χρήση των όπλων αυτών, δεν θα είχαμε σταματήσει να σκεφτόμαστε τον αντίκτυπο μιας ενδεχόμενης ε, στρατιωτικής παρέμβασης. Πολλά από τα ερωτήματα τα οποία είχα στο κεφάλι μου όταν μπήκα εδώ στην αίθουσα έχουν επιληθεί, αλλά και αυτό που είπε ο κ. Ντανζάν για, τα... για τις κυρώσεις. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από το διεθνές δίκαιο, θεωρώ. Εσείς τι θεωρείτε και ποια θα μπορούσε να είναι μια σχετική απόφαση για το θέμα αυτό. Και μια συγκεκριμένη ερώτηση να σας κάνω. Μια μελέτη της εταιρεία EIS, της ε, εταιρεία Συμβούλου για θέματα στρατιωτικά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ομάδες σχετικές με την Αλκάιντα αποτελούν την πλειονότητα των ανταρτών. Τα χρήματα και τα όπλα των Από πού προέρχονται. Μιλάμε για τη μείωση του εξοπλισμού. Αυτό ασφαλώς θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα πρέπει να αποτρέψουμε επιπλέον εξοπλισμό. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να συμβαίνει αυτό. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό θα ξέρουμε, πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά. και φυσικά το ρόλο της Ρωσίας, το οποίο, τον οποίο αναφέρατε και εσείς. Θα μπορούσε να ασκήσει πίεση η Ρωσία στον Ασάντ, πραγματική πίεση. Και αυτό θα είχε νόημα. Αλλά αυτό θα σήμαινε ότι η Δύση θα έπρεπε με τη σειρά της να ασκήσει πίεση στους αντάρτες. Μιλήστε μας γι' αυτό. Πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί. Θα μπορούσε. Καν να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Και θα εφαρμοστεί, θεωρείτε. Ευχαριστώ. Κύριε Λανσμπέργκης τώρα έχει το λόγο. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου κάποιες παρατηρήσεις που απασχολούν τον κόσμο η καταστροφή των χημικών θα πρέπει να συνοδεύεται με την καταστροφή, με την εξόντωση αυτών των εγκληματιών, των φωνιάδων, των εγκληματιών κατά της ανθρωπότητας, οπότε θα πρέπει να δούμε ότι αυτό έχει προτεραιότητα και όχι τίποτε άλλο. Ο κύριος Άσαντ θα τη γλιτώσει υπό την προστασία της Ρωσίας. ενθαρρύνεται στην επιθετική του στάση και όσον αφορά τη χρήση των χημικών ουσιαστικά. Το σαρίν έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκε. Άρα, θα έπρεπε το συντομότερο δυνατόν να του αποστερήσουμε τη χρήση των ε, χημικών, μια που δεν έχει καμία υπεύθυνη στάση. Μίλαμε τώρα για φόνο αμάχων, παιδιών, ανηλίκων. Επομένως, η λογική λέει ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα νέο ειδικό δικαστήριο για τα εγκλήματα της ανθρωπότητας στη Χάγη. Και να υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και να υπάρχουν κάποια αποτελέσματα ατράνταχτα όσον αφορά τις καταδίκες και, έτσι να ε, συνεχιστεί και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν κάποιο είδου έρευνα ε, που να οδηγεί σε αυτή την ε, αντιμετώπιση δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ και θα πρέπει να είσαστε συγκεκριμένοι και σύντομοι σε ερωτήσει σα. Ο κύριο Ζέμκε και η κυρία Αναγκόμε τελευταία. Ζέμκε. Χωρίς μικρόφωνο, κύριο Ζέμκε. Σας e, e, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω κάτι να συνεχίσω. Πάνω σε αυτό που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε, τα δύο συγκεκριμένα ζητήματα δηλαδή, όσον αφορά ε, την ε, ε, απομάκρυνση και την καταστροφή των χημικών. Η Συρία γνωρίζει ότι αυτά θα και ε, καταστραφούν τελικά. Και γι' αυτό και σας ερωτώ, Τι τέχνασμα θα χρησιμοποιήσουν τόσο ώστε να μην αποστηρθούν των χημικών. Μήπως ε, θα τα κρύψουν κάπου εκτός ε, επικρατείας τους. Ιδίως τα μικρότερα από αυτά τα όπλα. Μικρότερο βελληνικό. Μπάς και τα πάνε να τα κρύψουν στο Λίβανο ή στο Ιράν. Λέτε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. Δεύτερη ερώτηση. Συζητούμε για τα χημικά. Αλλά δεν φύγουμε τα βιολογικά όπλα. Μήπως επειδή μέχρι τώρα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή επειδή έχουμε πιστεί ότι η Συρία δεν έχει βιολογικά όπλα, γιατί δεν το συζητάμε. Για μένα μου φαίνεται περίεργο το, το, το, ότι υπάρχει τελείως μια σιωπή γύρω από αυτά τα όπλα, τα βιολογικά. Ξέρετε κάτι. Για να Χωρίς μικρόφωνο. Λέτε ότι τώρα θα ξεκινήσει ε, κάτι, κάτι σαν το παιχνίδι που κράτησε χρόνια με το Σαντάμ, δηλαδή σαν το ποντικό με τη γάτα, όσον αφορά τώρα δηλαδή για την καταστροφή των χημικών. Επίσης, όσον αφορά τη Ρωσία. Όσο περισσότερο ακούω για την ε, σύγκρουση αυτή, τόσο περισσότερο πείθομαι ότι έχουμε, εκτός από αυτόν τον πόλεμο, την, την αντιπαράθεση Ρωσίας Δύσης και Σιητών Σουνιτών. Αυτό δεν μπορούμε να το κρύβουμε. η προφητεία έχει γίνει η κατηγορία της Ρωσίας ότι η αντιπολίτευση είναι τρομοκράτες. Τι λέτε. Από πού προέκυψαν οι προτάσεις των Ρώσων. Πολλοί λένε ότι από τους Αμερικάνους ξεκίνησε. Σικόρσκι. Ήταν και θέμα βέβαια περιθωρίου ελιγμών από πλευρά Ομπάμα. Δεν είχε τόσο μεγάλο περιθώριο ελιγμών στο Κογκρέσο. Αλλά βέβαια κανένας δεν ε, ξεσκέπασε την πλόφα των ε, Ρώσων. Στον ΟΗΕ τι γίνεται. Τι, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε. Ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Και είναι και η Τουρκία βέβαια αλλά έχουμε και τους υποστηρικτές του, του, του κόλπου, της χώρας του κόλπου. Βέβαια και η Τουρκία είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα. Για πέστε μας. Τι λέτε για το ρόλο της ε, Τουρκίας, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα με τους ε, Κούρδους, αυτοί που έρχονται συνέχεια στο Ιράκ. Υπάρχουν και κάποιες αντιφάσεις. Έχουμε και το ΠΚΚ, το κουρδικό. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσει, τέλος. Ε, ιδίως όσον αφορά το Ιράν και τη Ρωσία που θα κάτσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε κάποιους παραγωγούς στη δικαιοσύνη του Άσαντ και των άλλων εγκληματιών στο δικαστήριο της Χάγης. Μήπως αυτό είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαν να κάνει οι διεθνείς κοινότητες. Δεν είναι αυτό το λιγότερο που μπορεί να γίνει όσον αφορά το ότι έχει απεμπολίσει την ευθύνη του ο Άσαντ για την προστασία του λαού του. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο ψήφισμα από κάπου. Πιέζει ο χρόνος, λέω ο Πρόεδρος. Εσείς έχετε το λόγο. Για να δούμε, να μην παραλείψω καμιά ερώτηση, τι θα γίνει με τα χημικά, πώς θα χτυπήσουμε τις συγκαταστάσεις. Σαφώς προέκυψε ότι τα σχετικά εργοστάσια δεν μπορούμε να τα χτυπήσουμε. Θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. θα λυθεί η ατμόσφαιρα ή κάποιοι ακραίοι θα μπορούσαν να τα ε, πάρουν. Πρέπει να έχουμε ίσως κάποιο είδους ε, αντικίνητρα για τη χρήση τους. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι θετική συνεργασία ή παρουσία για τα χημικά. Τώρα για το κατά πόσο αυτά μπορούν να πάνε να τα κρύψουν στο Ιράν ή στο Ρελίβανο, δεν το νομίζω. Δεν νομίζω ότι η Δύση θα επιτρέψει να κρυφτούν εκεί που είπατε τα χημικά στο λίγο της Χεσμπολάχ για παράδειγμα. Για τον εξοπλισμό τώρα, ναι, έχουν σημαντικά όπλα και τα περισσότερα προέρχονται από την Τουρκία και από τα κράτη του κόλπου. Κάποια λίγα και από την Ευρώπη. Αυτά για τους ε, αντάρτες. Δεν έχουν βαριά όπλα πάντως. Αντιαρματικά, ή ε, ε, αντιεροπορικά, γιατί υπήρξε ο φόβος ότι αν τους τα δώσουμε θα καταλήξουμε σε εξτρεμιστές. Το θέμα δεν είναι ότι χρειάζονται πιο βαριά όπλα. Και έτσι να υπάρξουν λιγότεροι θάνατοι. Απλώς. Το θέμα είναι ότι από πλευράς εξοπλισμού είναι ισχυρότατος ο Άσαντ και ποτέ δεν θα μπορέσουν να τον φτάσουν όσον αφορά τον εξοπλισμό ή τις αντιπολίτευσης. Ο σχετισμός των δυνάμεων είναι πολύ εις βάρος της αντιπολίτευσης. Δεν είναι θέμα το αν θα τους δώσουμε μερικά αντιαεροπορικά και μερικά αντιαρματικά. Αυτό είναι ψευδοεπιχείρημα. Μεγάλη υπεροχή της ε, κυβέρνησης. Χρειάζεται να δώσουμε πάρα πολλά όπλα για να αντισταθμίσουμε αυτή τη διαφορά. Το Κατάρα, η Αραβία αλλά και η Τουρκία βέβαια εξοπλίζουν. Και από ιδιώτες υπάρχει και χρηματοδότηση. Πολλά από τα χρήματα πάνε σε εξτρεμιστές. Κατάρ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, από εκεί προέρχονται. Από ιδιώτες ή από κρατικούς φορείς. Από τέτοια χρήματα. Δεν προσέχουν τόσο πολύ σε ποιον θα πάνε τα χρήματα όσο το ότι ο καθένας προσπαθεί να ε, προστατεύσει τα συμφέροντά του στην περιοχή. Αν τώρα τις ερώτηση για την Τουρκία. Δεν ξέρω γιατί σχέση με την Αλνάστρα, αλλά πάντως όντως στέλνουν χρήματα, όπλα και θα έπρεπε να ελέγχει περισσότερο η τουρκική κυβέρνηση. Και στη Βόρεια Συρία οι εξτρεμιστές έχουν ενισχυθεί πολύ. Δεν τους στηρίζει άμεσα η Τουρκία, αλλά πάντως από απλά συνόρων υπάρχει χαλαρότητα. Όλοι θα έχουν συμφέρον ε, να σταματήσουν τον Άσαντ με τα χημικά, γιατί ε, υπάρχει διάδοση τέτοιων όπλων. Και η Ρωσία επομένω θα πρέπει να προσέξει το πόσο υποστηρίζει έμεσα τη χρήση των χημικών. Αυτό όσον αφορά την Ρωσία, τι κόκκινε γραμμέ τη, το θέμα μου δεν είναι τι γίνεται με τον Ασάντ, είναι το τι γίνεται με την διεθνή ένωμη τάξη, τι γίνεται με τη ΣΥΒΑ. Αυτά όσον αφορά τον Κέρι και τη συμφωνία που αναγνώρισε την, τον ρόλο των Ρώσων. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για μονομερή επέμβαση της δύση. Άρα, δεν είναι θέμα διαδικασία. Είναι το πώς οι Ρώσοι δεν θα πιστεύουν ότι τους χειραγωγεί η Δύση. Το θέμα δεν είναι τι θα κάνει η, η Δύση, αλλά το πώς θα πιεστεί ο Άσαντ. Η Ρωσία, όπως είναι τώρα τα πράγματα, διευκολύνεται να τον υποστηρίξει τον Άσαντ. Και ξεκινάμε μια πολιτική διαδικασία σήμερα με την οποία είναι συνομιλητής ο Άσαντ. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος διαπραγμάτευσης. Οι Ιρανοί επίσης θα αποκτούν υπομόχλιο, θέλουν και αυτοί να υπασπιστούν τα συμφέροντά τους. Άρα έτσι πρέπει να ενεργήσουμε με, εξυπνάδα. Για τους κινδύνους τώρα ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το να μην επιτευχθεί διεθνής συμφωνία. Τίποτα πλευρά ΟΗΕ, τίποτα πλευρά Συμβουλίου Ασφαλείας, να μην βγει, οπότε να καταρρεύσουν οι προσπάθειες. Για μένα το θέμα είναι η, ο αφοπλισμός. Δεν βλέπω γρήγορα να ευωδώνεται. Είναι φίλος πόλεμος και τα πράγματα είναι δύσκολα. Δύο χρόνια πέρασαν, χωρίς ψήφισμα του ΟΗΕ, με διχασμό εθνικό, άρα. θα πρέπει με κάθε τρόπο να σταματήσει αυτού του είδους η σύγκρουση. Γιατί έχει ευρύτερη σημασία για κινδύνους. Να, ποιος είναι ο κίνδυνος. Να καταρρεύσουν οι προσπάθειες για συμφωνία. Και είπα, εάν ο Σαντάμ ξεφύγει από τους κανόνες, μπορεί να προχωρήσει μονομερός και εκτός ΙΕ. Πρόσφατα ήμουν στην Μόσχα και πάρα πολλοί διπλωμάτες ήταν εκεί και οι δύο Ευρωπαίοι λέγανε ότι η συμφωνία της Γενέβης μεταξύ Λαυρόφ και Κέρι προέβλεπε ότι το ψήφισμα του 7ου κεφαλαίου θα είναι δεύτερη φάση. Δεν θα προβλέπεται στο αρχικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οπότε οι Ρώσοι εδώ νομιμοποιούνται κάπως να πούνε ότι η Δύση προσπαθεί να πλασάρει σε πρώτη φάση το 7ο κεφάλαιο Εάν αλλάξουν τα δεδομένα, έτσι κι πρέπει να εμπλέξουμε και τη Ρωσία στις διπλωματεύσεις. Για τη λογοδοσία, για την τιμωρία που πρέπει να επιβληθεί στον Άσαντ, βεβαίω υπάρχει εδώ πέρα μια ηθική επιταγή. Να σταματήσει ο κόσμος να σκοτώνεται. Και άρα να μπει φρένο σε αυτή την κατάσταση που θα μπορούσε να πάει παντού, θα μπορούσε να έχει συνέπειες. Και όσον αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εάν κανείς ε, θεωρεί θα πρέπει να δώσει λόγο ο Ασάντ, ε, θα πρέπει κάπως να ακολουθήσει αυτό κάποιες διπλωματεύσεις. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε για δικαστήριο. Πρώτα πρέπει να προχωρήσει η πολιτική διαδικασία. Όλοι να πιέσουν όπου μπορούν για να κάτσουν όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. και. Θα βάλω τελεία. Και θα επανέλθουμε στις υπόλοιπες ερωτήσεις μετά, αλλά θα στον παρακαθήμενο θα δώσω τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Να προσπαθήσω να, να ομοτοποιήσω τις απαντήσεις. Καταρχάς, να πω ότι συμφωνώ με διάφορα από τα σχόλια που ακούστηκαν από τους βουλευτές σε σχέση με το πόσο σχετικά είναι τα χημικά όπλα στην όλη σφαγή που έχει λάβει η χώρα. Είναι μικρό το τμήμα των θανάτων. Μιλάμε ε, για τον ίδιο αριθμό ε, θανάτων όπως και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σήμερα στη Συρία και όπως και στην διαμάχη Ιρακράν. Ωστόσο, κάτι που δεν θα πρέπει να υποτιμάει ο κόσμος είναι η σημασία των χημικών όπλων για την ασφάλεια γενικότερα στην Συρία. Μου προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι είχε η Συρία χημικά όπλα τακτικής ε, φύσης, γιατί ως τώρα το χημικό οπλοστάσιο της Συρίας θεωρείται στρατηγική σημασίας, παρόμοια με τα πυρηνικά όπλα της, του Ισραήλ. Είναι κρυμμένα, κανείς δεν τα συζητάει, όλοι ξέρουν ότι υπάρχουν και χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση που η χώρα η ίδια αντιμετωπίσει κίνδυνο για την ύπαρξή της. Έτσι όπως εξελίσσεται ο πόλεμος, μιλάμε για μία απειλή της ύπαρξης της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν η χώρα τα τελευταία δύο χρόνια η Συρία έχει αρχίσει να αναπτύσσει τέτοια τακτική φύσεω όπλα, ίσως και γι' αυτό να ήταν τόσο αυθαίρετη η χρήση τους. Για τον Ασάντ, με άλλα λόγια, ίσως τίθεται θέμα του κατά πόσον θα επιζήσει τον πόλεμο αυτό και αυτές οι πιθανότητες είναι αρκετά περιορισμένες. Η Ντάλλος θα μπορέσει να, ενδεχομένως να υπάρξει κλιμάκωση στο άμεσο μέλλον για την ε, καταστροφή των όπλων χημικής καταστροφής. Σε διάφορους τρόπους μπορούμε να εξετάσουμε, όπως είπα και στην παρουσίασή μου, δεν ξέρω ακόμα τι θα αποφασίσει το εκτελεστικό συμβούλιο του OPCOW. Είναι απόφαση δικιά του. και ενδεχομένως να αλλάξουν και οι ημερομηνίε στόχος για την ε, συμφωνία βάσει των τεχνικών αναλύσεων των ε, καταστάσεων επιτόπου. Δεν θέλω λοιπόν να εικάσω γι' αυτό. Κοιτώντα τις εμπειρίες στο Ιράκ την δεκαετία του 90, κάποιες μεθοδολογίες καταστροφής ήταν για παράδειγμα να χυθούν οι Δραστικέ ουσίε στην έρημο, στην άμμο. Τώρα το κατά πόσο κάτι τέτοιο θα ήταν ε, αποτελεσματικό σήμερα δεν ξέρω, είναι άλλο θέμα, αλλά ήταν αποτελεσματικό να θαυτούν στη γη. Ε, έκρηξη στο ε, υπέδαφος, καύση των χημικών όπλων, ελεγχόμενη ωστόσο. Θα πρέπει κανείς φυσικά να λάβει υπόψη και τις παράγωγες ουσίες σε περίπτωση που υπάρχει αέρας για παράδειγμα υπάρχουν ε, κάποιες κινητές εγκαταστάσεις τις έχουν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες η Γερμανία, η Σουηδία για παράδειγμα εξ όσων γνωρίζω που χρησιμοποιούνται για την ε, καταστροφή ε, βιομηχανικών τοξικών υλών και η ΙΠΑ και η Ιαπωνία έχει τέτοια, έχουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Πόσες τέτοιες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να μεταφερθούν άμεσα στη Συρία. Όλα αυτά είναι στοιχεία που θα πρέπει να λεφτούν υπόψη. Το να γίνει, να γίνει επίθεση για να καταστραφούν τα χημικά όπλα, αυτό δεν θα το σύστηνα. Γιατί θα κάναμε ακριβώς αυτό που προσπαθούμε να αποφύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση τα όπλα ιδιαίτερα αν βρίσκονται αποθηκευμένα σε κάποιο ανοιχτό χώρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταστραφούν όλες αυτές οι ουσίες, θα δημιουργηθούν νέφη τα οποία θα κινηθούν προς αστικές ε, περιοχές. Να θυμηθείτε και κάποιες ασθένειες ε, μετά τον πόλεμο του κόλπου που σχετίζονταν με τέτοιες καταστροφές ε, ουσιών μετά το κουβέιτ για το ρόλο της Ρωσίας. Ο μεγαλύτερος ρόλος έγκυται στην διπλωματία. Δεν χρειάζεται να υποστηρίζουμε τον Πούτιν ή και το τρέχον πολιτικό σύστημα στη Ρωσία για να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για μια ευκαιρία την οποία θα πρέπει να δράξουμε. Δεν νομίζω όμως ότι επειδή κάποιος ε, αν δράτει μια ευκαιρία θα πρέπει εκ των προτέρων να τον ε, καταδικάσουμε επειδή δεν μας αρέσει το καθεστώς ή το συγκεκριμένο άτομο. Έχουν γίνει τεράστια στρατηγικά σφάλματα και πολλά εξ αυτών ε, στην Δύση. Καταρχάς τον Αύγουστο του περσινού έτους ο πρόεδρος Ομπάμα ε, εξέδωσε μια ανακοίνωση και ανέφερε ποια ήταν οι κόκκινες γραμμές του και έτσι στριμώχθηκε στη γωνία γιατί ουσιαστικά κάλεσε οποιονδήποτε είχε χημικά όπλα να ελέγξει πού ήταν αυτές οι κόκκινες γραμμές και πώς θα μπορούσε να τις προσπεράσει. Μία άλλη γκάφα που έγινε. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία και σε κάποιο βαθμό και οι Ηνωμένε Πολιτείε εστιάστηκαν στα θύματα των χημικών όπλων γιατί αυτό ξεκίνησε ένα ολόκληρο διάλογο για ανθρωπιστικά ζητήματα, για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πάρα πολύ σημαντικά μεν, αλλά φυσικά μέσα αντιμετωπίζουμε το θέμα του πώς κάποιοι εκατοντάδες ε, νεκρών συγκρίνονται με χιλιάδες εκατοντάδες νεκρούς. Και γιατί δεν έχουμε επέμβει σε μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις. Άρα εδώ πέρα έχουμε λίγο κολλήσει τον τοίχο. Η κατάσταση λοιπόν σήμερα πώς διαμορφώνεται. Ξέρω ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου προσπαθούμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλειας βάσει αξιών, δημιουργείται το πρόβλημα της δικαιοσύνης για τα θύματα, οι λίγες εκατοντάδες που σκοτώθηκαν, και του αφοπλισμού, το οποίο έχει να κάνει με το πόσο υποφέρει ο κόσμος και να κοιτάξουμε όμως και τις μακρο, μακροοικονομικές ε, συνέπειες. Αυτό όμως σημαίνει ο αφοπλισμός. Και κοιτώντας τι σημαίνει λοιπόν η έννοια του αφοπλισμού, θα, θα διαπιστώσουμε ότι σε οποιαδήποτε συνθήκη και συμφωνία αφοπλισμού πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ως ίσο τον εταίρο του. Ιδάλλως δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγματεύσεων και συνομιλιών. Και θεωρώ ότι αυτή η ευκαιρία που ξαφνικά αναδύθηκε από το χάος της αντίθεσης αυτής ανθρωπινών δικαιωμάτων κατά χημικών όπλων δημιουργεί διάφορες ευκαιρίες και συμφωνώ με τον Τζούλιεν ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία αλλά μπορεί να είναι πάρα πολύ ε, για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ας την αδράξουμε λοιπόν. Δίνει σύμφωνη, δίνει κάποια νομιμότητα στον Ασάντ και στο όλο θέμα. Αλλά ίσως γι' αυτό το λόγο ακριβώς υπάρχει και μία υποψία ελπίδας για να υπάρξει μια διαπραγμάτευση που θα μας κάνει να βγούμε από τον πόλεμο, ακριβώς γιατί θα αναγνωριστεί. Δεν θα αμφισβητηθεί, δεν θα εξαφανιστεί στις διαπραγματεύσεις αυτές το καθεστώ του και ο ίδιος. Θα, υπάρξει, θα είναι λοιπόν ένα μέλος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τα χημικά όπλα στο πλουστάσιο του Σαντ είναι για να επιβιώσει το καθεστώς και το κράτος. Αυτό που Κάποιος ανέφερε το Άνσκομπ στο, στην δεκαετία του 90 και στο Ιράκ. Η κατάσταση ήταν διαφορετική από πολλές απόψεις. Δεν, ήταν, δεν υπήρχε πόλεμος. Αλλά το ψήφισμα 687 του Συμβουλίου Ασφαλείας ουσιαστικά επιβλήθηκε σε μια ευτυμένη, σαν μέρος. Ο Σαντάμ λοιπόν είχε κάθε λόγο να αποφύγει τον εντοπισμό των χημικών όπλων γιατί ό,τι μπορούσε να κρύψει για κάποιους ε, μήνες, ε, για κάποιο χρόνο έστω, μπορούσε να το διατηρήσει για μελλοντική χρήση. Αλλά στη Συρία και στο Ιράκ μπορεί να υπάρχει η εξής ως προς τις εξελίξεις. Αν στο Ιράκ τελικά δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Αυτό οφειλόταν γιατί έγινε μια ε, μετάβαση από την αφοπλισμό στην, ε, στο αίτημα για αλλαγή καθεστώτος. Άρα, ενώ αρχικά δεν υπήρχε κίνητρο για τον Χουσέι να συνεργαστεί, σε μετέπειτα στάδιο δεν είχε κίνητρο να συνεργαστεί, γιατί ουσιαστικά ήθελαν να τον ξεφροντωθούν. Το είδαμε λοιπόν και με την ε, εισβολή στο Ιράκ το 2003 επειδή υποτίθεται ότι είχε χημικά όπλα. Δεν λέω ότι από εσά εξαρτάται η πολιτική απόφαση για το ποιε είναι οι προτεραιότητε. Απλά λέω ότι από πλευρά αφοπλισμού παρουσιάζονται κάποιε ευκαιρίε για να επιληθεί ο πόλεμο, να επιληθεί το θέμα των μη συμβατικών όπλων στη Μέση Ανατολή. Είναι πραγματικά ίχνος ελπίδα. Δεν είναι σαφέ αν υπάρχει η ελπίδα αυτή, αλλά πραγματικά εξετάστε και αυτή τη λύση. Μπορούν να καταστραφούν όλα τα χημικά όπλα στην Συρία. Είναι δύσκολη ερώτηση. Ωστόσο, να έχουμε υπόψη ότι πρόκειται για μια διαδικασία. Το βασικό το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι το εξής. Η Συρία στις 14 Οκτωβρίου θα προσυπογράψει πλήρως ε, τη συνθήκη για τα χημικά όπλα. Το είπα ότι η συνθήκη αφοπλισμού είναι συνεργατική ασφάλεια. Συνεργατική με βάση σαφείς υποχρεώσεις. Και ενώ σε πολλές ε, χώρες ενδεχομένως να υπάρχει οπλοστάσια, μπορεί να προκύψουν ε, περαιτέρω ε, συμφωνίες αφοπλισμού. Ο EPCW δεν πρόκειται να καταστρέψει τα όπλα. Είναι υπεύθυνο για να επιβλέψει την ε, καταστροφή των όπλων. Αυτό θα πρέπει να πιστοποιήσετε. Έχουν καταστραφεί τα όπλα. Οι επιχειρήσεις τώρα καταστροφής και η ευθύνη είναι στη Συρία. Αλλά επειδή η Συρία θα είναι τμήμα της σύμβασης όπως έγινε και στην Αλβανία, όπως έγινε και σε άλλες χώρες, θα υπάρξει διεθνής αρρωγή. Η Λιβύη, η ΙΠΑ, η Γερμανία και διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν δηλώσει ήδη ότι πρόκειται να διαθέσουν και πόρους και εμπριογνώμονες. Τώρα η μεταφορά των χημικών όπλων στο Ιράν και στο Λίβανο σε καμία περίπτωση ούτε που να το σκεφτείτε. Το Ιράν είναι μέλος της Σύμβασης των Χημικών Όπλων θα ήταν τεράστια παραβίαση για μια χώρα που έχει υποστεί τεράστιες απώλειες επί 8 χρόνια από χημικά όπλα και γνωρίζει ακριβώς τι γνωρίζει, τι σημαίνει όταν ότι η διεθνής κοινότητα δεν θέλει να βοηθήσει ακόμη και όταν κανείς έχει τόσα πολλά θύματα. Είναι εταίρος της Συρίας μάλιστα, αλλά το Ιράν θα βοηθήσει σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις και την εφαρμογή της συνθήκης. Το ίδιο ισχύει και για τη Ρωσία. Ο Λίβανος δεν είναι λύση και ο Λίβανος είναι μέρος ε, της συνθήκης. Μόνο το Ισραήλ από όλες τις γειτονικές χώρες δεν είναι μέλος της συνθήκης αυτής. Αλλά όταν ο Λίβανος επικύρωσε τη σύμβαση, η Χεσμολά ήταν μέρος της κυβέρνησης. Η Χεσμολά έχει δεσμευτεί πολιτικά για να τηρήσει την συνθήκη και επανελειμμένα το έχει τονίσει αυτό έκτοτε. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι οι κινήσεις αυτές είναι πραγματικά πιστευτά σενάρια σε ό,τι αφορά τα χημικά όπλα, σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές ικανότητες Χρειάζονται, ξέρετε, μεγάλες ποσότητες προκειμένου να υπάρχει στρατηγική, στρατιωτική εφαρμογή, εκτός και αν μιλάμε για μικρού τύπου τέτοια όπλα. Τελευταίο θέμα. Κάποιος έθεσε το θέμα των βιολογικών όπλων στη Συρία. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα τέτοιο επίθεση στη Συρία. Κάποιες, μάλλον καμία χώρα στην παρούσα φάση δεν ε, παραδέχεται να κατέχει τέτοια βιολογικά όπλα. Ωστόσο, αυτό που μου δίνει κάποια βεβαιότητα ήταν η συνέντευξη του Ασάντ στο Σπίγκελ, στο πρακτικό Σπίγκελ, τον Ιανουάριο του 2009 όταν τον ρώτησαν για τις ικανότητες και το δυναμικό μη συμβητικών όπλων, κυρίως σε ό,τι αφορά πρινικά όπλα και σε σχέση με το πλωστάσιο του Ισραήλ. Τον ρώτησαν λοιπόν για τα πυρηνικά και τα βιολογικά όπλα και είπε ότι όχι, όχι, τίποτα. Για τα χημικά όπλα η αυθόρμητη αντίδρασή του ήταν «Α, κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι διαφορετικό». Δεν ήταν και καλυμμένη η απάντησή του. Ήταν σχετικά ειλικρινής. Μπορεί λοιπόν η Συρία να έχει ένα πρόγραμμα αμυντικό, όπως έχουν και πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει κάτι το επιθετικό cette Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση για τη Συρία. Οι δύο παρεμβάσεις σας επέτρεψαν να έχουμε πολύ συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία. Ε, βέβαια, το είπα εξ αρχής ότι δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλο το πρόβλημα, να λύσουμε το Συριακό αλλά εν πάση περιπτώσει ε, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση δεν είναι απίθανο να ξαναδιοργανώσουμε τέτοιου είδους ε, συνεδρίες. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ τα πέντε λεπτά που μας μένουν για να για να σας αναφέρω τα όσα έγιναν στην περασμένη εβδομάδα στην επίσκεψη που κάναμε ε, στο Ταλίν, στην Εστονία. Μια επίσκεψη που στόχο είχε καταρχήν να επισκεφθούμε το κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ για την κυβερνοάμυνα και το εκμεταλλευτήκαμε για να συναντήσουμε τους εστονούς ε, βουλευτές καθώς και τον Υπουργό Αμήνης. Σύντομη επίσκεψη, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με το κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ. Μπορέσαμε να ακούσουμε πολύ ε, περιστατωμένες εισηγήσεις για τις έρευνες που γίνονται εκεί και που οδήγησαν στη δημοσίευση δύο αρκετά ενδιαφερόντων έργων, διότι για μας τους ευρωβουλευτές είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα μάλιστα, γιατί αναφέρονται στο νομικό πλαίσιο της κυβερνοάμυνας και της κυβερνοασφάλειας ε, και είναι πραγματικά ένα τομέας στον οποίο Υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία ορισμών, διατάξεων, ερμηνεών, αναχώρα, αναοργανισμό, που η προσπάθεια που γίνεται στο Ταλίν για να εξορθολογισμό του νομικού πλαισίου για αυτές τις δράσεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και Είχαμε και επαφές με τους ε, ομολόγους μας, βουλευτές της Επιτροπής Αμήνης του Κοινοβουλίου της Εστονίας και μετά και με τον Υπουργό Αμήνης και ανταλλάξαμε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για το ποιες μπορεί να είναι η, ποια μπορεί να είναι η συνεννόηση για μια μικρή χώρα τις οποίες ε, οι θρεπτικές ε, οι ένοπλες δυνάμεις είναι περιορισμένες, αλλά συμμετέχουν στις αποστολές του ΝΑΤΟ. Σημαντική ήταν η συμμετοχή των εστονικών δυνάμεων στην αποστολή ISAF στο Αφγανιστάν με απώλειες που αναλογικά με την ανάπτυξη των στρατευμάτων ήταν μεγάλες. Μια ανάπτυξη που μας ανέφερε στη... και για την αποστολή στο Μουαλή ε, ο Υπουργός. Πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε, αλλά και πρώτη προτεραιότητα και απόλυτη προτεραιότητα που στρέφεται προς τους Ρώσους γείτονες. Μία στάση και ένας λόγος αρκετά επιθετικός που ε, ε, ανησυχεί πολλούς βεβαίως στην Εστονία αλλά και άλλες χώρες της περιοχής που δεν θα πρέπει να την προσιοποιήσουμε. Νομίζω λοιπόν πως ήταν αυτές οι επισκέψεις σε χώρες που δεν είναι απαραίτητα οι χώρες που θεωρούμε αυθόρμητα ως σημαντικούς πυλώνες της ΚΕΠΑ, δεδομένου του μικρού μεγέθου των ενόπλων δυνάμεών τους, ωστόσο μας επιτρέπουν να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα της αμυντικής προσπάθειας μιας τέτοιας χώρας, μικρής χώρας και έπειτα την ανησυχία που για την συλλογική άμυνα που είναι πρώτη προτεραιότητα και εξάλλου και η βασική μέρημνα μιας αμυντικής πολιτικής. Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η συνάντηση. Βρήκαμε συνομιλητές πολύ ενήμερους για τα θέματα αυτά και για την ΚΕΠΑ θα πρέπει να πω, αν και προτεραιότητα δίνεται στο ΝΑΤΟ όσον αφορά την συλλογική άμυνα πράγμα που είναι απόλυτα κατανοητό. Πάντως διαπίστωσα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Και προσθέτω και κλείνω ότι σε αυτές τις μετακινήσεις είναι πολύ καλό να συμμετέχουν δραστήρια οι εστονοί συνάδελφοι της υποεπιτροπής. Πρώτος ε, και καλύτερος ο κ. Κέλλαμ που είναι εδώ, ο κ. Στάραντ και η κυρία Όγιουλαντ ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τις αρχές της Εστονίας να κατανοήσουν ότι οι ευρωβουλευτές οι Εστονοί είναι δραστήριοι στις επιτροπές μας, στην Υποεπιτροπή Αμήνης και στην Επιτροπή Εξωτερικών. Και γι' αυτό και ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά να, να συμμετέχουμε σε αυτήν την αποστολή. Κύριε Κέλλα, μου θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που δώσατε για επίσκεψη στις εγκαταστάσεις αυτές να ευχαριστήσω και τον αντιπρόεδρο μας, από τον Κύπριο αντιπρόεδρό μας που συμμετείχε. Νομίζω και βεβαίως είναι καλά τα νέα ότι η Γαλλία θα γίνει θα συμβάλλει πλήρως, θα γίνει πλήρης ε, ε, συνεισφέρουν στο, στο, στο κέντρο αριστείας. Ε, να πω όμως στο, στο κολέγιο που έχουμε στο Τόρτο, που είναι το τρίτο αγγλόφωνο κολέγιο τέτοιου τύπου στην Ευρώπη, ε, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σε λιγότερο από 10 χρόνια το κολέγιο μας αυτό ε, είδε χίλιους φοιτητές που δεν προέρχονται μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Βοσνία, Ουκρανία, τις ε, δημοκρατίες ε, πέρα από τον Κάφκασο, Μακεδονία, Μολδαβία, Κροατία και ένα σωρό άλλες χώρες. Θα μπορούσε δηλαδή να πει κανείς ότι εδώ έχουμε pooling and sharing στην πράξη. Και αυτό αποτελεί μια πολύ καλή βάση για προσωπικές σχέσεις και κοινέ αξίες. Και επίσης μας είπαν οι συνάδελφοι από το Κολέγιο Βαλτικής Άμυνας. Το βασικό τους πρόβλημα είναι πώς θα μοιραστούν τους ανθρώπινους πόρους, ε, ε, γιατί χρειάζονται σε διάφορα μέρη ταυτόχρονα. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε την αλληλεγγύη στην πράξη, σε δράση, διότι όπως ανέφερε και ο συνάδελφος Λαντσμπέργη σήμερα, το ΝΑΤΟ δεν θεωρεί πως η ασφάλειά μας απειλείται από τα ανατολικά μας, και, από τα ανατολικά μας σήμερα, αλλά κάποιες χώρες που βρήνε στα ανατολικά μας σήμερα θεωρούν εμάς ως εχθρούς. Και αυτά λοιπόν πρέπει πολύ σοβαρά να τα εξετάσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν θέλει κανείς άλλο να πάρει το λόγο. Ε, είμαστε ακριβώς στην ώρα μας. Σας ευχαριστώ ε, και καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Όχι. Στις 14 Οκτωβρίου θα συνεδριάσουμε εκ νέου. Ε, ακυρώσαμε τη σύνοδο της επόμενης 3ης Οκτωβρίου, για τη θεωρήσαμε ότι το ποσοστό συμμετοχής θα ήταν ε, μικρό. Γι' αυτό προτιμήσαμε να το αναβάλουμε για μια άλλη ημερομηνία. Θα γίνει συνεδρίαση λοιπόν στις 14 Οκτωβρίου η επόμενη.